Okay. Uh, now we will... Θα συνεχίσουμε τώρα ε, με την κανονική συνεδρίαση της Επιτροπής Γιούρη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων. Δεν θέλω να σας πετάξω έξω από την αίθουσα, αλλά θα ήθελα να αποχωρήσετε όμως όσοι δεν είστε σχετικοί. In the meantime, we με το μεταξύ να εγκρίνουμε τα πρακτικά. Έρχομαι λοιπόν στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για τα πρακτικά. Βλέπω πως όχι. Αυτό σημαίνει ότι τα πρακτικά ε, της συνεδρίασης της 11 η Ιανουαρίου του 2016 εγκρίνονται. Επομένως, τώρα έχουμε μείνει μεταξύ μας. Κυρίως, υπάρχει μια εξαίρεση, αλλά μπορούμε να συνεχίσουμε με την εξέταση του σημείου 5 της ημερησίας διάταξης. Εξέταση του εγγράφου εργασίας για την προστασία των ευπαθών ανηλίκων, ενηλίκων, ενηλίκων να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ζωέλ Μπερζεγού. Πριν το κάνω όμως, να σας πω ότι είναι μια πρόταση ίδιας πρωτοβουλίας που ακολουθεί ε, τη δουλειά του Λόπες ε, Ιστουρίθ στην ε, κυρία ε, Μπερζερό, η νομική προστασία των ευάλωτων ενηλίκων αφορά άτομα άνω των 18 ετών που προσωρινά ή μονίμως είναι ανίκανα να διαχειριστούν την περιουσία τους ή το άτομο τους. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι ο καθένας μας είναι δυνάμει ευάλωτος ενήλικας και μπορεί άμεσα ή άμεσα να επηρεαστεί από το πρόβλημα αυτό γιατί αυτή η τροτότητα μπορεί να έχει σωματικό ή ψυχικό χαρακτήρα, μπορεί να οφείλεται σε ένα τυχημα ή απλώς να είναι απόρρια βία νευροεκφυλιστικής ασθένεια ή ε, της προχωρημένης ηλικίας. Στη Γαλλία δυστυχώς είχαμε διάσημες περιπτώσεις τέτοιων ευάλωτων ατόμων που προβλήθηκαν ιδιαίτερα στην δημοσιότητα. Δεν ξέρω, ε, για παράδειγμα την κυρία Λιλιάν Μπετανκούρ ή Βενσάν Λαμπέρ, δεν ξέρω αν είχαν την ίδια πύχηση και σε εσά. Ήταν πλούσιοι διάσημοι άνθρωποι που ακριβώς επειδή ήταν απομονωμένοι πολλοί τους εκμεταλλεύτηκαν. Ο κύριος Λαμπέρ ήταν νέος, έπαθε ατύχημα και έχασε την ικανότητα να μπορεί να διχειρίσει τη ζωή του. Ε, ε, οι ηλικιωμένοι υπερήλικες ε, είναι όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη ε, της παράτασης του προσδόκιμου ζωής. Έχουμε όλο και περισσότερους λοιπόν ευάλωτους ενήλικες και αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα πραγματικό νομικό πρόβλημα. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί ένα από τα θεμέλια θεμελιώδης λήθους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ε, οι άνθρωποι θα πρέπει να διακινούνται και να μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δημιουργεί διασυνοριακούς ε, νομικούς δεσμούς ανάλογα με το που βρίσκεται η περιουσία ή ο τόπος διαμονής που μπορεί να βρίσκεται στην αλλοδαπή ή λόγω ε, σύναψη συνδικής σχέσης με αλλοδαπό. Βέβαια, ή ε, επίσης αγορά ακινήτου σε χώρα με πιο το κλίμα. Και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους. Γιατί έχουμε πολλού ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν διασυνοριακού τέτοιου νομικού δεσμού. Για παράδειγμα, οι βοηθοί μα, οι ε, ευρωϊπάλληλοι που είναι υποχρεωμένοι να διαμένουν στο Βέλγιο. Τι θα συμβεί αν το κάποιο πάθει ατύχημα ή αρρωστήσει και καταστεί ανίκανο να διαχειριστεί την περιουσία του και τη ζωή του ποια νομοθεσία θα εφαρμοστεί, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο, ποια είναι η αρμόδια δικαιοδοσία, ποιος ε, ε, θα είναι ο δικαστικός τους εκπρόσωπος ή θα ασχοληθεί με τη φροντίδα τους. Και αν ε, κάποιος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί στο Βέλγιο θα ισχύσουν αυτόματα και στην πατρίδα του ή στη νέα χώρα διαμονής. Θα πρέπει να ξεκινήσουν νέες νομικές διαδικασίες για να αναγνωριστούν όλα αυτά τα μέτρα ή να υπάρξει μια συμμόρφωση ή να ανανεωθούν. Πολλά ζητήματα λοιπόν που αφορούν τους ευάλωτους ενήλικες. Θα πρέπει να βρεθούν σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν τέτοιες ξεκάθαρες απαντήσεις γιατί δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα συνεκτικό και κατάλληλο νομοθετικό πλέγμα για τους ευάλωτους ενήλικες. Τα συστήματα προστασίας των κρατών μελών διαφέρουν δυστυχώς μεταξύ τους. Και δεν είναι και πολύ ρεαλιστικό τη στιγμή αυτή να προτείνουμε μία εναρμόνιση των ε, διαφόρων ενόμων συστημάτων εξαιτία του μεγάλου κατακαιρματισμού και των τεραστίων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ του. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα προστασίας με μέτρα που θα αντιμετωπίζουν ε, αποτελεσματικά αυτόν τον ευάλωτο χαρακτήρα. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε ένα ψήφισμα ζητώντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα, ε, μια νομοθετική πρόταση προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών ε, προκειμένου να βελτιωθεί η αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων για ευάλωτους ενήλικες. Μέχρι στιγμής όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει υποβάλει καμία τέτοια νομοθετική πρόταση. Σας προτείνω ένα έγγραφο εργασίας που προς το παρόν αποτελεί μόνο μια βάση για τη συζήτηση και γι' αυτό θα ήθελα τα σχόλια, τις απόψεις και τη συνεργασία σας. Μέχρι στιγμής ε, το μόνο νομοθετικό μέσο που έχουμε για τις διασυνοριακές ε, διαφορές για τα ευάλωτα άτομα είναι η Σύμβαση της Χάγης της 13ης Ιανουαρίου του 2000. 20 περίπου χώρες την έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής, 8 μόνο την έχουν επικυρώσει. Η Γερμανία, η Αυστρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, μόνο για την Σκοτία, η Φιλανδία, η Τσεχία, η Εστονία και η Γαλλία. Και πολύ πρόσφατα το πριγκεπάτο του Μόνακο. Δυστυχώς δεν επαρκεί αυτή η χαμηλή επικύρωση για την ε, εφαρμογή της προτάσεις μας, οι συστάσεις μας είναι εξή. Επίγει και καλό θα ήταν να, να ενθαρρύνουμε κάποιους ελάχιστους παρανομαστές. Να επικυρωθεί η σύμβαση της Χάγης που προβλέπει ένα ισορροπημένο, σαφές, συνεκτικό και ευκρινές σύστημα. Πέραν όμως των ενθαρρύνσεων αυτών που μπορεί να είναι και μάζες γιατί ε, για μερικές χώρες μέλη θα, απαιτήσει προηγουμένως ε, δικαστική νομική μεταρρύθμιση, κάτι που είναι και δαπανηρό και χρονοβόρο, γιατί πρόσφατα είχαμε στη Γαλλία μια τέτοια μεταρρύθμιση και το κόστος ήταν τεράστιο. Γιατί εγώ έχω επαφή ε, με ευάλωτα άτομα και μάλιστα ένας βοηθός μου ήταν εντολέας μιας τέτοιας, εντολοδόχος μιας τέτοιας ε, περίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε την εφαρμογή της Σύμβασης τη Χάγης που διευκολύνει την αναγνώριση εκτέλεση αποφάσεων για ευάλωτα άτομα που τη χάνουν ε, και αποφελούνται από μέτρα προστασίας. Ε, επίσης, λόγω των χαρακτηριστικών αυτού του προβλήματος θα προτιμούσαμε κανονισμό αντί για οδηγία, παρόλο που γνωρίζω ότι αυτό είναι ευσεβής περισσότερο. Τέλος, ένα σημείο που κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί αφορά την οτροπία. Είναι σημαντικό, αν θέλουμε να λάβουμε υπόψη την ελευθερία και την αξιοπρέπεια του κάθε ατόμου, να το λάβουμε υπόψη. Με βάση τη σύμβαση της Χάγης ε, ε, αφορά την εντολή ανικανότητας. Εμείς έχουμε εντολή για μελλοντική προστασία που είναι κάτι παρεφερέ στη Γαλλία και ξεκίνησε το 2007 με τη νέα μεταρρύθμιση. Οπότε ο καθένα που έχει ε, ικανότητα δικαιοπραξίας μπορεί να ε, διαλέξει, προβλέποντας για μια μελλοντική ανικανότητα, έναν ή δύο ε, ε, ανθρώπους που θα αναβάλουν την περιουσία και τον άτομό του. Και φυσικά θα ξεκινήσει η ισχύ αυτή τη εντολής μόνο σε περίπτωση αλλίωσης της ικανότητας σωματικής ή πνευματικής αυτού του ατόμου. Επίσης, είναι σημαντικό να γίνει σεβαστή αυτή η βούληση. Βέβαια, κάτι τέτοιο ίσως μας φέρει ε, σε δύσκολη θέση γιατί ε, μας φέρνει αντιμέτωπου με ένα δύσκολο πρόβλημα που είναι η απώλεια των ε, ικανοτήτων μας. Το θέμα όμως είναι ότι με μια τέτοια πρόταση δεν υφίσταται απλώς κανείς τα μέτρα προστασίας αλλά μπορεί να τα επιλέξει με τρόπο που γίνονται σεβαστές η ελευθερία και η αξιοπρέπειά του. Θα πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε την αναγνώριση και την εφαρμογή τέτοιας εντολής από τα κράτη-μέλη χωρίς να χρειαστούν νέες διαδικασίες. Ε, κάνοντας σεβαστή την βούληση ε, του μελλοντικά ανίκανου ευάλωτου ατόμου. Επίσης θα πρέπει να λυθεί και το θέμα των διασυνοριακών κληρονομικών διαδοχών. Δεν είναι αρκετό για να επιλυθεί το ζήτημα των ευάλωτων ατόμων. Θα πρέπει επιτέλους με νυφάλιο τρόπο και πριν φτάσουμε σε διαδικασία του κατεπήγοντος, κάτι που δεν θα αργήσει, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Thank you very much, Mr. Kester. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Κέστερ. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Θα ήθελα να σχολιάσω το εξής. Μιλούμε για την ε, ευαλωτότητα των ηλικιωμένων, αλλά πρέπει να δούμε το θέμα και ε, στα πλαίσια της, δημογρα... της δημογραφικής αλλαγής των κοινωνιών μας. Αν δούμε τις δικές μας κοινωνίες, αυτό, αυτές χαρακτηρίζονται από το ότι τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια μεγάλη αύξηση υπερηλίκων. Και ακριβώς οι άνθρωποι αυτοί είναι, έχουν αυξημένο ποσοστό ευαλωτότητας, ευαισθησίας και στην Ευρώπη έχουμε μια κατάσταση όπου αυτοί οι υπερήλικες ε, πρέπει να μπουν σε κάποιους ε, οίκους ευγυρίας όπου ουσιαστικά η ε, ελευθερία τους δεν την χάνει κανένα σεβασμού. Οπότε αυτό, αυτή την πτυχή ίσως θα έπρεπε να την τονίσουμε λίγο περισσότερο. Πώς μπορούμε δηλαδή στην Ευρώπη να έχουμε ένα ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο ώστε ακριβώς τα δικαιώματα των υπερηλίκων που είτε πνευματικά είτε σωματικά είναι αδύναμοι, να μπορούμε να, διατηρήσουμε, να τα διατηρήσουμε και σε τέτοιους οίκους ευγυρίας, αν αυτοί χρειάζεται να νοσηλευτούν σε αυτούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νεγκρέσκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με την εισηγήτρια. Πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτή την κατάσταση των ευάλωτων ατόμων. Αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κάτι αντίστοιχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν είχε γίνει τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Δεν έχει γίνει τίποτα ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής αυτών των ατόμων. Έχουμε κάποια προβλήματα σε σχέση ακριβώ με τα ως, ε, με τα ως ενήλικες ε, σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε έναν ορισμό αλλά η ερμηνεία που δίνεται στον ορισμό από τα διάφορα κράτη-μέλη δεν είναι η ίδια. Και πρέπει, νομίζω, να βρεθεί μία κοινή ερμηνεία στον ορισμό που έχουμε. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό, έχουμε και κάποιους σχετικούς συναφείς όρους ε, και έννοιες ε, ε, όπως η αξιολόγηση των πνευματικών δυνατοτήτων των ατόμων αυτών που επίσης ορίζονται με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη και πρέπει και αυτό να το αναγνωρίσουμε και στην έκθεση αυτή να προσπαθήσουμε να ζητήσουμε την ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών για τον καθορισμό του ορισμού αυτών των σημαντικών όρων. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι λόγω του ότι δεν έχουμε ορισμό συγκεκριμένο, αυτό σημαίνει έξτρα κόστος για τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα πρέπει να τονιστεί, γιατί καμιά φορά όταν ε, συζητούμε για όρους, για ερμηνείες κτλ, τίνουμε να ξεχνούμε ότι ε, πέραν του προβλήματος που δημιουργεί η έλλειψή τους, δημιουργεί και έξτρα κόστος Οπότε αυτό νομίζω ότι θα μπορούσαμε να το τονίσουμε για να πιέσουμε τα κρατημέλη να συνεργαστούν πιο στενά και να δημιουργήσουν ένα κοινό πλαίσιο όρων για όλους αυτούς τους και μια κοινή, ένα κοινό πλαίσιο ερμηνεών για όλους αυτούς τους όρους. Επίσης, κάτι άλλο που θέλω να τονίσω είναι ότι είναι σαφές ε, και για μένα και για τη συνάδελφο ότι θα πρέπει να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση ώστε νομικώς να προστατεύσουμε τους ευαίσθητους ενήλικες, τους ευάλωτους ενήλικες. αν θα τους πούμε τώρα, ε, αν θα μιλούμε για ηλικιωμένους, αν θα μιλούμε για άτομα με αναπηρία, αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες χρειάζονται προστασία και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θα πρέπει να βελτιώσει αυτή ακριβώς την προστασία που τους παρέχεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κομοντίνη. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ την εισηγήτρια για το πολύ καλό έγγραφο που προετοίμασε. Έχω κάποια σχόλια που θέλω να μοιραστώ μαζί σας με βάση το έγγραφο εργασία που έχουμε στα χέρια μας. Είναι προφανές ότι ένα κοινό σύστημα που προστατεύει τους ε, ευάλωτους ε, ενήλικες όπου η ε, ζωή τους βρίσκεται σε διάφορα κράτη-μέλη όντως χρειάζεται προστασία και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούν να ασκήσουν όλα τους τα πολιτικά και θεμελιώδη δικαιώματα. Συχνά η κατάσταση αυτή αφορά Στου ε, ηλικιωμένου που αποφασίζουν να συνταξιδοτηθούν σε ένα άλλο κράτος μέλος ή θέλουν να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό βεβαίω έχει να κάνει με μεγάλου κίνδυνου, με υψηλότερο κίνδυνο ασθένεια, που σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο για την ύπαρξη κάποια ευαισθησία. Πρέπει βεβαίως να δούμε τι σημαίνει ευαισθησία ή ευαλωτότητα και να θέσουμε κάποια όρια στο πεδίο εφαρμογή ε, και στη δουλειά που θα κάνουμε. Γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιο ε, έχει ανικανότητα δικαιοπραξία κατά ανάγκη αν, είναι, αν θεωρείται ευάλωτο ενήλικα. Μπορεί να θέλει όντω να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα. Ε, οπότε σε τέτοιε περιπτώσει πρέπει να δούμε ποιο είναι ο ορισμό και ποιο είναι το πεδίο που θέλουμε να δουλέψουμε. Θέλουμε να έχουμε μια εναρμονισμένη, ε, εναρμονισμένο ορισμό ή θέλουμε να έχουμε ένα σύστημα που παρέχει μόνο προστασία σε αυτούς που θεωρούνται ε, ανίκανοι λιγοπραξίας επειδή βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος ή όταν βρίσκονται σε ένα κράτος μέλος ή ακόμα και στην χώρα καταγωγής τους όταν θέλουν να εξασκήσουν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης που έχουν. Νομίζω ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που έχουμε στην έκθεση αυτή είναι οι διαφορέ που υπάρχουν ήδη μεταξύ των κρατών μελών. Στην δουλειά μα λοιπόν πρέπει να καταγράψουμε τα διάφορα συστήματα που υφίστανται στι ένωμες τάξει των κρατών μελών και να δούμε πού είναι τα όρια μα και πού θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια μα. Για παράδειγμα, κάποια κράτη-μέλη δεν παράσχουν ούτε αναγνωρίζουν ε, την αξιοδότηση των ε, νομικών για άτομα που θέλουν να ονομάσουν κάποιον ως ε, προστάτη τους. Ε, αυτοί, αυτά τα άτομα μπορεί να πρέπει να πάρουν απόφαση για ε, κάποια ιατρική θεραπεία σε περίπτωση που οι, τα άτομα αυτά έχουν πάθει κάποιο ατύχημα ή ασθένεια και ε, κυρίως όταν υπάρχει περίπτωση όπου αρνούνται την λήψη θεραπείας. Και υπάρχουν και δυστυχώς διαφορετικές ε, βάσεις ε, για την κατάργηση αυτών των διαδικασιών σε περίπτωση που τα άτομα αυτά δεν επιθυμούν κάτι παρόμοιο. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μία λύση για να καλυφθούν όλες αυτές οι διαφορές, γιατί αυτές οι διαφορές έχουν να κάνουν κυρίως με, την, με θέματα όταν, όπου τα άτομα αυτά θέλουν να διατηρήσουν τις, ε, τα δικαιώματα που έχουν, Εκτός όμως αν υπάρχουν κάποιες πράξεις οι οποίες αναγνωρίζονται μέσα στα κρατημέλη αλλά θεωρούνται ότι είναι αντίθετες με την δημόσια αυτή πολιτική. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί ε, όταν κάποια άτομα μπορεί να, πρέπει να λάβουν απόφαση για την θεραπεία που θα λάβουν μετά από κάποιο ατύχημα ή για πράξεις που δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς και που μπορούμε να τις ε, καταγράψουμε και να τις ρυθμίσουμε ε, βάζοντας κάποιες ε, ελάχιστες απαιτήσεις ή ελάχιστες διαδικασίες για να υπάρξει αναγνώριση των νομικών πράξεων που μπορεί να διεξαχθούν σε άλλε, που να εκτελεστούν σε άλλο κράτο μέλο με το οποίο μπορεί να έχει κάποια σχέση το άτομο αυτό και βεβαίω να υπάρχουν κανόνε για αμοιβαία εμπιστοσύνη για τι διάφορε διαδικασίε των κρατών μελών ώστε να ε, διευκολυνθεί αυτή η αναγνώριση. Η συγκίτρια νομίζω ότι σωστά καταγράφει την, ε, την, ε, την σύμβαση τη Χάγη όπου αναφέρονται όλα αυτά τα θέματα για να υπάρξει βελτίωση της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων σε όλα τα κράτη κρατη κυρίω, ε, επειδή τα περισσοτερα κρατημέλη δεν έχουν επικυρώσει ή υπογράψει αυτή την σύμβαση. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα όσα προτείνει η υπογράψη αυτη αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η σύμβαση αυτή έχει ε, καταφέρει να αποφευθούν ε, διαμάχε μεταξύ των νομικών συστημάτων σε περίπτωση αρμοδιότητα και ε, υπάρχουν φυσικά θέματα όπου πρέπει να προσπαθήσουμε ακριβώς να αποφύγουμε τέτοιου είδους διαμάχες ε, ακριβώς για να προστατεύσουμε τους ευάλωτους ε, ενήλικες. Πρέπει να έχουμε κοινέ ελάχιστες αρχές για να, με βάση τα όσα υπάρχουν στα συστήματα των κρατών μελών πριν, όμως έχουμε ένα συγκεκριμένο ε, νομικό μέσο, είτε κανονισμό είτε οδηγία, θα πρέπει να είναι σαφή τα θέματα που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Είναι λοιπόν σημαντική όλη αυτή η διαδικασία που θα διευκολύνει την ε, ελευθερία διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίω εγώ θα συνεργαστώ στενά με την εισηγήτρια και με του υπόλοιπου εισηγητέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Λεμπρετών παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο να προστατεύουμε τους ευάλωτους ενήλικες και μάλιστα με διασωνοριακή προστασία. Και η έκθεση αυτή πράγματι ασχολείται με αυτό το θέμα και γι' αυτό αξίζει που υπάρχει. Ωστόσο δεν συμφωνώ με το συμπέρασμά της. Η λογική λύση είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη να επικυρώσουν τη σύμβαση της Χάγης του 2000, ένα κείμενο υψηλής ποιότητας, διότι ορίζει την αρμόδια δικαιοδοσία που είναι ε, ε, η δικαιοδοσία του κράτους όπου έχει τη συνήθη κατοικία του ενδιαφερόμενος και προβλέπει συγκεκριμένες διατάξεις προστασίας όπως είναι η ε, εντολή ανικανότητας λήψης αποφάσεων το 2007 έχουμε ένα σχετικό νομικό εργαλείο στη Γαλλία και μπορώ και εγώ να σχολιάσω το γαλλικό σύστημα. Είναι ένα εξαιρετικό σύστημα και σας προτείνω να ξαναδιαβάσετε τη σύμβαση της Χάγης και να εμπνευστείτε από αυτήν. Ενθαρρύνω τα κρατημέλη να την επικυρώσουν. Ωστόσο, δεν συμφωνώ με την ύπαρξη ευρωπαϊκού κανονισμού, ούτε καν ευρωπαϊκής οδηγίας για το θέμα αυτό. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα και θα πρέπει να σεβαστούμε το περιθώριο ελιγμό των κρατών μελών, δηλαδή την εθνική τους κυριαρχία. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω την παρέμβασή τους ε, εκφράζοντας την έκπλησή μου για το οικονομικό επιχείρημα της έκθεσης. Μας λέτε ότι 16 εκατομμύρια το χρόνο στοιχίζει η απουσία ε, νομικής διάταξης για το θέμα αυτό στο ενωσιακό δίκαιο. Εγώ νομίζω ότι είναι ε, εκτός τόπου και χρόνο αυτό που λέτε γιατί είναι το θέμα εξαιρετικά πολιτικό και σε καμία περίπτωση οικονομικό. Ο κύριος Ντιουγάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να μιλήσω κι εγώ στα γαλλικά. Χαίρομαι που παίρνω το λόγο μετά τον κύριο Λεμπρετό. Γιατί γιατί όχι μόνο προφανώς αλλά κυρίως φυσικά και δεν συμμερίζομαι την άποψή του και θα ήθελα να εκφράσω την πλήρη μου στήριξη στη δουλειά της κυρίας Μπερσεγό. Δεν θα μακρηγορήσω, γιατί σύμφωνα απόλυτος με την έκθεση αυτή, αντιθέτως με τον κύριο Λεμπρετό, πιστεύω ότι πρέπει να πάμε προς μια εναρμόνιση, προς κοινή ε, νομοθετική ρύθμιση είτε με τη μορφή του κανονισμού είτε με τη μορφή της οδηγίας γιατί φτάνουμε στον πυρήνα της κοινωνικής Ευρώπης της υπεράσπισης των πιο αδύναμων και αυτό είναι μία από τις αποστολές της Ευρώπης η οποία δυστυχώς την έχει κάπως ξεχάσει δίνοντας προβάδισμα στα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα και δίνοντας το προβάδισμα στις οικονομικές δυνάμεις. Έτσι, ε, σφυριλατούμε την καρδιά της Ευρώπης και πραγματικά το, χρειάζονται, το χρειάζεται αυτό η Ευρώπη. Και παίρνω το λόγο για να εκφράσω την πλήρη μου στήριξη στην κυρία Μπερζέγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελούκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, την, την εισηγητριά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνεισηγήτρια, έλεγα, για την ε, πολύ περιεκτική αυτή έκθεση, η οποία απεικονίζει τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της έλλειψης διασυνοριακής συνεργασίας για το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη λύση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008, κάτι το οποίο έλαβε υπόψη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην όλη τη δουλειά μέχρι και σήμερα. Και θα ήθελα να ε, υπενθυμίσω ότι το ψήφισμα του 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ε, γνωμοδότηση ίδιας πρωτοβουλίας μόλις έχει υπάρξει επαρκής εμπειρία από την εφαρμογή της σύμβασης της Χάγης και αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Ανέκαθεν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλούσε τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση, να την επικυρώσουν και να μπορέσει έτσι να παρακολουθήσει την εφαρμογή της. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι ήδη από το 2010 αλλά και το, στη συνέχεια το 2014 και το 2015 έχουμε διανύμει ερωτηματολόγιο στο Συμβούλιο, στα κράτη-μέλη με διάφορες ερωτήσεις αναφορικά με την εφαρμογή στην πράξη της Σύμβασης της Χάγης του 2000. Του 2000. Τουλάχιστον απευθυνόμενη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα κράτη-μέλη που πράγματι ε, κύρωσαν τη Σύμβαση και απευθύναμε ερωτήματα στα λοιπά κράτη-μέλη γιατί δεν το έχουν πράξει αυτό. Και όλη αυτή τη διαβούλευση την έχουμε ε, διαβιβάσει στην εισηγήτρια. Από όλη αυτή τη διαβούλευση φαίνεται ότι τα, ε, τα κράτη-μέλη τη μου ελετούν την δυνατότητα κύρωσης της Σύμβασης της Χάγης και όσο κράτη-μέλη την κύρωσαν θεωρούν ότι είναι πολύ καλή και θεωρούν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι μέχρι σήμερα είχαν χρειαστεί να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά ελάχιστες περιπτώσεις. Στη Γαλλία για παράδειγμα 24 περιπτώσεις μόνο, στη Γερμανία 21, στη Σκοτία μία μόνο περίπτωση. Είναι σαφές λοιπόν ότι ε, με τόσο λίγα δεδομένα μια νομοθετική πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν στοιχειοθετείται επαρκώς, δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη ύπαρξης νομοθετικής πρωτοβουλίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα έχουμε συγχρηματοδοτήσει τη διαδικτυακή τοποθεσία, το, το, την ιστοσελίδα του Συμβουλίου των Συμβολεογράφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του δικτύου αυτού notaries. Επίσης έχουμε ε, διαδώσει την Εθνική Νομοθεσία για το θέμα αυτό και φέτος θα μεταφράσουμε το επεξηγηματικό υπόμνημα στη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων. Θα το μεταφράσουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες εκτός από τα αγγλικά και τα γαλλικά που είναι οι επίσημες γλώσσες της διάσκεψης ε, της Χάγης ε, για την ε, σύνταξη της Σύμβασης της Χάγης και στην Ομάδα Εργασίας για θέματα αστικού δικαίου στο Συμβούλιο θα ζητήσουμε την άποψη των κρατών μελών ξανά. Θα κάνουμε έναν απολογισμό των εξελίξεων κατά τη διάρκεια του 2015 και θα δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η κύρωση της Σύμβασης της Χάγης και ποιες είναι οι νέες περιπτώσεις που χρειάστηκε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια του 2015. Επομένως, θα ήθελα να καθησυχάσω την εισηγήτρια λέγοντάς της ότι παρακολουθούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Την 1η Πρώτου του 2009 τέθηκε η σύμβαση σε ισχύ. Είναι μια νέα σύμβαση Και δεδομένου του γεγονός ότι λίγες χώρες την έχουν κυρώσει, όπως ε, σας είπα ήδη, δεν υπάρχει επαρκής εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει και τον τρόπο με τον οποίο έχει εφαρμοστεί. Όμως, ε, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας τη θεωρούν πολύ καλή και θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να την κυρώσουν. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε και θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο ε, να δούμε δηλαδή κατά πόσο υπάρχουν πιο αυστηροί τρόποι θα έλεγα να ε, τα κράτη-μέλη να ανεβάσουν ταχύτητα, να επιταχύνουν τη διαδικασία κύρωσης της σύμβασης. Σας ευχαριστώ κυρία Μπερσεγόν για τις καταληκτικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ όλους τους παρεμβαίνοντες και ευχαριστώ κυρίως τον κύριο Ντιουγάν, ο οποίος πράγματι μίλησε ε, για την ουσία του προβλήματος. Η Ευρώπη δημιουργήθηκε για να πλουστεύσει τη ζωή των πολιτών και όχι να την περιπλέξει. Ε, συνήθως υπάρχουν κανονισμοί που περιπλέκουν τη ζωή των πολιτών και εδώ έχουμε ένα νόμο που θα διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων που δεν μπορούν να αυτοδιαχειριστούν οι ίδιοι. Και είναι σημαντικό η Ευρώπη να υιοθετήσει τέτοιου είδους νομοθεσία. Δεν είναι καθόλου πολιτικό το ζήτημα. Ε, σε αυτού του είδους την νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Αντιθέτως, ο, ανεξαρτήτως πολιτικών ιδεών και τάσεων θα πρέπει όλοι να βρούμε μια κοινή συνισταμένη για να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Και πράγματι πρέπει να βρεθεί ένας ε, ορισμός αποδεκτός ε, τουλάχιστον στο ίσον ε, σημείο του για το τι εστί ποιος είναι ευάλωτος άνθρωπος. Στη Γαλλία υπάρχουν τρόποι να διαχειριστούν ε, την ε, περιουσία τους μέχρι ότου τεθούν υπό επιτροπή, υπό κυδαιμονία. Μπορεί δηλαδή κανείς να ορίσει ε, όταν έχει ο ίδιος ήδη καλή υγεία και σώστας φρένας να ορίσει έναν άλλον άνθρωπο που εκεί τη βουλήσει ο οποίος θα διαχειριστεί τα περιουσιακά του όταν ο πρώτος δεν θα είναι σε θέση να παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό του. Ε, η σύμβαση της Χάγης είναι εξαιρετικό εργαλείο. Το πρόβλημα είναι ότι κανένα κράτος δεν την κυρώνει. Μόνο 8 κράτη-μέλη την έχουν κυρώσει. Και την περασμένη εβδομάδα με την κυρία Χαουτάλα ήμουνα στη Χάγη, ε, είδα τους ανθρώπους εκεί, και φοβούνται ότι το ενωσιακό δίκαιο θα αποδυναμώσει τη δική τους ε, διεθνή ε, συνθήκη, σύμβαση. Τι θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε να είμαστε ε, στα απόνερα μιας διεθνούς διάσκεψης όπως ήταν η διάσκεψη για τη Σύμβαση της Χάγης ή θέλουμε να έχουμε πρωτογενές δικό μας ενωσιακό δίκαιο. Και γιατί υπάρχουν τόσες λίγες περιπτώσεις. Π.χ. όταν ένας Άγγλος ζει στη Γαλλία θα σας πω γιατί είναι τόσο λίγες περιπτώσεις. Όταν γίνεται ευάλωτος και επιστρέφει ε, στην πατρίδα του, κανείς δεν το ξέρει εκεί. Έχουμε έναν οργανισμό στη Γαλλία που ε, ασχολείται με τα ευάλωτα άτομα και αυτός ο οργανισμός δεν ενημερώνει κανέναν. Ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρουν καθόλου καμία δημόσια διοίκηση, καμίας χώρας. Τους αφήνουμε ελεύθερους και τέλος. Και δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτούς δεν μπορεί κανείς να διαχειριστεί ανθρώπινα όντα από τον ε, τελευταίο όροφο του ψηλού κτηρίου στο οποίο δουλεύει. Αντιθέτως πρέπει να κατέβει επί να τους δει από κοντά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λόγω της ευαλωτότητάς τους κινδυνεύουν. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το σημείο 5 και περνάμε στο σημείο 6. Το σημείο 6 προβλέπει εξέταση του εγγράφου εργασίας με θέμα τη θέσπιση ελάχιστων κοινών προτύπων για την πολιτική δικονομία. Πρόκειται για ένα θέμα που ενδιαφέρει και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου και μάλιστα η Επιτροπή μας έχει θέσει παρατηρητή στο ELI, ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δικαίου και θα δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή μας για το θέμα αυτό, στον κύριο Εμίλ Ράντζεφ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω το έγγραφο εργασίας μου με θέμα τη θέσπιση ελάχιστων κοινών προτύπων για την πολιτική δικονομία. Στόχος του εγγράφου είναι να κάνει μια επισκόπηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε θέματα δικονομικού δικαίου. Όπως ξέρετε, η κατάργηση του εκτελεστήριου τίτλου Εξεκουάτορ διευκόλυνε την ελεύθερη διακίνηση των δικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών, αλλά αυτό καθιστά την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών ιδιαίτερα σημαντική. Από νομική άποψη πάντως, η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαστικών αρχών σημαίνει ότι τα εθνικά δικαιικά συστήματα μεταξύ των κρατών μελών ακολουθούν παρόμοιους οικονομικούς κανόνες για να εξασφαλίσουν δίκαιες δίκες σε θέματα αστικού δικαίου. Η εμπιστοσύνη επιτείνει την ασφάλεια δικαίου και ταυτόχρονα προβλέπει τη δέουσα σταθερότητα και προβλεψιμότητα για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έγγραφο εργασία μου πραγματοποιεί μια ανάλυση των νομοθετικών ε, ε, όρων για μια μελλοντική έκθεση πρωτοβουλία προκειμένου να καταλήξουμε σε ελάχιστα πρότυπα δικονομικού δικαίου, πολιτικής δικονομίας. Μάλιστα, οι νομοθετικές επιλογές ε, στηρίζονται σε διαφορετικές νομικές βάσεις. Έχουμε δύο διατάξει στις στη συνθήκη που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις νομικές βάσεις για μια μελλοντική έκθεση. Για παράδειγμα, έχουμε τη γενική διάταξη του άρθρου 114 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρίνεται σκόπιμη για την ε, υιοθέτηση νομοθεσίας που αφορά και διασυνοριακές περιπτώσεις και εθνικές αρκεί τα μέτρα που θεσπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης υπάρχει ειδική διάταξη, το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρμοδιότητα να διευρύνει τη δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, αρκεί να έχουν ένα διασυνοριακό χαρακτήρα, διασυνοριακές συνέπειες. Στην περίπτωση αυτή, το διασυνοριακό στοιχείο, ο διασυνοριακός χαρακτήρας θα πρέπει να τύχει διασταλτική ερμηνεία και να μην θεωρείται ως συνώνυμο της, ε, του διακανονισμού διασυνοριακών διαφορών. Από την άλλη πλευρά μπορούμε να έχουμε και τομεακές ε, οδηγίες με βάση το άρθρο 114 ή τομεακά νομοθετικά μέσα. Έτσι μπορούμε να επηρεάσουμε κάποια στοιχεία της δικονομικής ε, διαδικασίας ε, σε κάποιες υποθέσεις αστικού δικαίου ή να επιλέξουμε κάποια οριζόντια νομικά μέσα για να εναρμονίσουμε τις εθνικές πολιτικές της σε περίπτωση που υπάρχουν διασυνοριακά στοιχεία ασχέτως τομέα. Επίσης έχουμε και κάποια προαιρετικά μέσα που θεσπίζουν μια σειρά δικονομικών κανόνων που εφαρμόζονται παράλληλα με τους εθνικούς. Τα μέσα εναρμόνισης ισχύουν για εθνικέ ε, δικονομικέ διατάξεις και υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να εναρμονίσουν τους εθνικούς τους κανόνες προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Υπάρχει θεωρητικά και μία τρίτη επιλογή. Μια και υπάρχει μία επικάλυψη μεταξύ των δύο άρθρων, το 81 και το 114, ε, στα θέματα εναρμόνισης της ε, πολιτικής οικονομίας που μπορεί να χρειάζεται για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά να ισχύει για διασυνοριακές περιπτώσεις. Βέβαια, εδώ χρειαζόταν μια διπλή νομική βάση. Καλό θα ήταν όμως να ζητήσουμε και τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ποια είναι η κατάλληλη νομική βάση για τέτοια θέματα θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε, να ζητήσουμε την γνωμοδότηση αυτή για την επόμενη μας συνεδρίαση. Και τώρα περιμένω την ε, άποψη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και φυσικά και τις δικές σας απόψεις και σχόλια. Η κυρία Διάννα Βόλι, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαίου, βρίσκεται εδώ σήμερα και χαίρομαι ιδιαίτερος για την παρουσία της. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα και πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να ακούσουμε την κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον συνάδελφο τον κύριο Ράντεφ ότι το έγγραφο είναι εξαιρετικής ποιότητας, πολύ αξιόλογο, γιατί πραγματικά κάνει μια επισκόπηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτικής οικονομίας. Και μετά την πρωινή ακρόση που είχαμε, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ των δικαιικών συστημάτων των κρατών μελών. Αν θέλουμε πραγματικά να υλοποιήσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων και μάλιστα με εύρυθμο τρόπο. Αυτή βέβαια η αμοιβαία εμπιστοσύνη δεν νοείται παρά μόνο όταν υπάρχει βεβαιότητα ότι τηρούνται και γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των διαδίκων σε όλα τα κράτη-μέλη. Δικαίωμα πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δικαίωμα υπεράσπιση, αλλά και μια σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των, των εναγόντων και των εναγωμένων. Βέβαια, η τήρηση όλων αυτών των αρχών γίνεται περίπλοκη. Υπάρχει το ζήτημα καταρχήν τη νομική βάση. Καθόλου εύκολο. Και ελπίζω η συζήτηση που θα κάνουμε να μας διαφωτίσει για τα θέματα της νομικής βάσης. Μάλιστα, η ρήτρα αυτοεξαίρεση ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη Ιρλανδία και τη Δανία ε, δεν διευκολύνουν ουδόλω αυτό το θέμα. Ποια είναι η κατάλληλη νομοθετική προσέγγιση, τα προαιρετικά νομικά μέσα, ε, οδηγίε οδηγίες με ελάχιστα πρότυπα, οριζόντιος ε, ε, τρόπος εναρμόνισης. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατή μια μέγιστη εναρμόνιση. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι καλή τύχη για να καταλήξουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Και χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί παρακολουθώ και συμμετέχω σε αυτό το θέμα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ρόζνερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που οργανώσατε την ανταλλαγή απόψεων για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα κοινά ελάχιστα πρότυπα πολιτικής δικονομίας και Καλωσορίζουμε βεβαίω και την ε, πλήρη ανάλυση που έγινε για το κείμενο που παρουσιάστηκε σήμερα για την πιθανή νομική βάση για ένα κείμενο που θα καλύπτει τι ε, αρχέ για την ε, κοινή πολιτική δικονομία. Ξέρουμε ότι τα θέματα αυτά είναι ιδιαίτερω σημαντικά όχι μόνο για το ποινικό αλλά και για το αστικό δίκαιο. Όταν υπάρχει άρνηση εκτέλεση ή αναγνώριση από κάποιο άλλο κράτο μέλο μια αστική απόφαση προκύπτει κυρίω από αμφιβολίε που υπάρχουν λόγω των διαφορετικών διαδικασιών που υπάρχουν στα αυτό λοιπόν είναι ε, σημείο πυρήνα για την ε, ύπαρξη αμοιβέ εμπιστοσύνη, που είναι ο πυρήνα ουσιαστικά της ε, καλής λειτουργίας του κοινού χώρου δικαιοσύνης ελευθερίας. Στην ανακοίνωση της Κομισιόν Δικαιοσύνη 2020 αναφέρεται αυτό ακριβώς το θέμα που μιλά για την παράδοση εγγράφων ε, την λήψη αποδεικτικών στοιχείων και την εξασφάλιση των, καλύτερων, των συμφερόντων του παιδιού σε αστικέ ε, διαδικασίε. Ε, αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν διαδικαστικούς κανόνες και θα αναφέρω τον κανονισμό για την παράδοση εγγράφων, την επίδοση εγγράφων και των αποδεικτικών στοιχείων, οι ευρωπαϊκές διαδικασίες για τις μικρές απαιτήσει, η ευρωπαϊκή εντολή πληρωμής, διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών και άλλοι διαδικαστικοί κανόνες που υπάρχουν σε πιο γενικά ε, αστικά εργαλεία όπως η Βρυξέλλες 1 ή η Βρυξέλλες 2α, οι σχετικοί κανονισμοί. Η νομική βάση που χρησιμοποιείται για αυτά τα εργαλεία ε, είναι το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς καμία εξαίρεση και ο προκάτοχός του στην Συνθήκη, στην συνθήκη Δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρθρο 65. Επίσης, ε, η ε, διαμεσολάβηση και οι νομικές ε, οδηγίες που προσπαθούν να λύσουν διάφορα προβλήματα σε αστικές διασυνοριακές υποθέσεις βασίζονται στο άρθρο 65 επίσης της συνθήκης. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σωστά στο έγγραφο εργασία που παρουσιάστηκε σήμερα, κάποια ατομιακή νομοθεσία περιλαμβάνει τέτοιες, τέτοιους κανόνες πολιτικής δικονομίας, όπως τα πνευματικά δικαιώματα και σχετική οδηγία ή η οδηγία ζημιών για το, από το αντιτράστ. Ε, αυτό το, στο άρθρο 1 και 14 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, τα, τα άρθρα 1 και 14 χρησιμοποιούνται ως νομική βάση. Βεβαίως θα πρέπει να δούμε και, τις, και τους υπόλοιπου κανόνε για την πολιτική δικονομία. Το εγγραφό πολύ σωστά αναφέρει ότι η πιο σωστή νομική βάση, η πιο κατάλληλη νομική βάση για μια μελλοντική παρέμβαση στον τομέα αυτό θα πρέπει να καθοριστεί ανάλογα με το συγκεκριμένο ε, περιεχόμενο που θα λάβει το σχετικό εργαλείο. Για το σκοπό λοιπόν αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, κάνει, έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις σε ό,τι αφορά την πολιτική δικονομία. Κάνουμε λοιπόν ε, μια ε, συνολική ε, συγκριτική ανάλυση των διαδικασιών στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να αναλύσουμε την σωστή εφαρμογή του σχετικού κανονισμού και να ορίσουμε κάποιους κανόνες που ίσως θα χρειάζονταν να δράσει ή παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για παράδειγμα, διασυνοριακή επίδοση εγγράφων θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς τους τομείς όπου η δυνατότητα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας θα μπορούσε να διερευνηθεί για να μειωθούν έτσι και τα μέτρα διαμεσολάβησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια νέα μελέτη για την εθνική πολιτική δικονομία. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης θα μας δείξουν κατά πόσο και σε ποιο βαθμό η υπάρχουσα απόκληση των ε, κανόνων σε εθνικό επίπεδο εμποδίζει την ε, πραγμάτωση των στόχων της ε, ελεύθερης διακίνησης των αποφάσεων, υπονομεύοντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Όντως θεωρούμε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εντατικοποίηση ή εκτέλεση των ε, ελάχιστων προτύπων στην πολιτική δικονομία θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό στην ε, διαφοροποίηση των ε, νομικών παραδόσεων των κρατών μελών και της νομοθεσίας τους και βεβαίως προς όφελος των νομικών και των φυσικών προσώπων. Ευχαριστώ. Thank you as well. Εγώ ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Οπότε να ακούσουμε τον κύριο Ραντεύ και πάλι, αν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για την ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέση της ε, για το ζήτημα αυτό. Ε, είδατε ότι μελετήσαμε τις απόψεις σας ε, όταν συντάσαμε την έκθεση αυτή και βεβαίως ε, ο καθορισμός αυτών των κοινών ελάχιστων προτύπων είναι μια δουλειά εν εξελίξη. Ελπίζω λοιπόν ότι όπως ξεκινήσαμε την διαδικασία αυτή θα δουλέψουμε όλοι αποτελεσματικά ώστε να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση. Βεβαίως ακόμη περιμένουμε την έκθεση που προετοιμάζεται για την προσθέμενη αξία από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το, την Άνοιξη θα γίνει ένα ε, εργαστήριο, ένα σεμινάριο για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι οι επιπλέον πληροφορίες που θα λάβουμε θα μας οδηγήσουν στο να καταλήξουμε σε ένα έγγραφο που θα μπορέσει να συντονίσει την πολιτική ε, δικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να διευκολύνονται και να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη, να υπάρχει πιο εύκολη αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων των διαφόρων κρατών μελών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τα ίσα ή ισότιμα δικαιώματα και τη δίκαιη δίκη για τους πολίτες μας. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κλείνουμε λοιπόν και το σημείο 6. Πάμε στο σημείο 7. Ανταλλαγή απόψεων μιας ε, πρότασης ε, ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας για την έκθεση διασυνορική αναγνώρισης των υιοθεσιών. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Σβιεύκα. <coughs> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάμε σε μια πιο ουσιαστική φάση των εργασιών επί της εκθέσεως με θέμα της διεθνής υιοθεσία. Στα τέλη του ε, προηγούμενου έτους, στις αρχές του Δεκεμβρίου, ε, διοργανώσαμε ένα εργαστήριο με θέμα την, τα διασυνοριακά νομικά ζητήματα των υιοθεσιών. Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το εργαστήριο ε, και μας διαφώτισε για τα πολύ σημαντικά αυτά θέματα και διαπιστώσαμε πόσο περίπλοκο και πόσο λεπτό και ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα που αφορά τις διαδικασίες υιοθεσίας, ε, τις διεθνείς υιοθεσίες συγκεκριμένα. Επίσης, είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η υιοθεσία δημιουργήθηκε για να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες για την ε, ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού. Αυτό ήταν ο γενεσιουργός της λόγος δεν έγινε υιοθεσία για να εξασφαλίσει ε, απογόνους σε γενείς που βιολογικά δεν μπορούσαν να έχουν δικά τους παιδιά. Σημαντικότερο δεν είναι το συμφέρον του παιδιού. Γι' αυτό δημιουργήθηκε η υιοθεσία. Και το ζητούμενο δεν είναι η ικανοποίηση των γονέων, αλλά των παιδιών. Αν και φαίνεται ότι στην πορεία έχει ανατραπεί κάπως αυτός ο στόχος. Θα πρέπει λοιπόν να επανέλθουμε στο γενεσιουργό λόγο, στον λόγο ύπαρξης της υιοθεσίας που είναι το συμφέρον των παιδιών. Οι εμπειρογνώμονες στο εργαστήριο που διοργανώσαμε μας παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα των προβλημάτων που οφείλονται στη διαφοροποίηση των εθνικών συστημάτων ε, που ισχύουν για την υιοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, μας επισήμαναν τα προβλήματα που προκύπτουν από τις διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών. Ήταν κρίμα που ήμασταν ε, λίγοι από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων ε, είχαμε πολύ περισσότερους από την Επιτροπή Αναφορών. Πάντως, ε, πολλά ε, υποθέσεις που ακούσαμε και πολλά ζητήματα που αναφέρθηκαν στην δημόσια αυτή στο εργοστήρι αυτό, θα αντικατοπτριστούν στην έκθεσή μου. Όπως σας είπα, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το θέμα των διεθνών νομοθεσιών. Γι' αυτό και θα ήθελα η έκθεσή μου να διαιρεθεί σε δύο τμήματα. Γιατί θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διαχωρίσουμε τις νομοθετικές στοιχές που αποτελούν αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις μη νομοθετικές πτυχές της διεθνούς ομοθεσίας γιατί έχουμε αρμοδιότητες που είναι εξαιρετικά σημαντικές και είναι απολύτως απαραίτητο να τις αναφέρουμε και να χαράξουμε το δρόμο για την επίλυση των προβλημάτων. Οπότε το πρώτο τμήμα της έκθεσής μου θα είναι νομοθετικό και θα αφιερωθεί αυτό το πρώτο νομοθετικό τμήμα της έκθεσης στην αναφορά του θέματος των εθνικών υιοθεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα αναφέρουμε την περίπτωση που είχαμε θεσία με βάση το εθνικό σύστημα και στη συνέχεια οι γονεί, μετά από κάποιο χρόνο αποφασίζουν να αλλάξουν τον τόπο διαμονή τους και μετακομίζουν σε άλλο κράτο μέλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και από τη στιγμή που έγινε μια εθνική νομοθεσία, αυτόματα αναγνωρίζεται και σε άλλο κράτος αυτή η νομοθεσία όπως συμβαίνει για υιοθεσίε που γίνονται με βάση την συνθήκη της, τη σύμβαση συγγνώμη, της Χάγης. Όπως όμως ήθιστε σε τέτοιου είδους καταστάσεις και εδώ έχουμε κάποια προβλήματα. Έχουμε προβλήματα που εμφανίζονται και που μας προβληματίζουν και αυτό θα πρέπει και να εγγύψουμε σε αυτά. Γιατί λοιπόν ανακύπτουν τα προβλήματα. Γιατί δεν έχουμε σήμερα και κατά πάσα πιθανότητα ποτέ δεν θα αποκτήσουμε έναν ενιαίο ορισμό της οικογένειας. Επίσης δεν έχουμε κοινή προσέγγιση, τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν έχουμε κοινή αντίληψη, κοινή προσέγγιση για τον ορισμό των ατόμων που ε, έχουν δικαίωμα να υιοθετήσουν παιδιά. Οπότε μία αυτόματη αναγνώριση της εθνικής νομοθεσίας είναι αδύνατη στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν διαρωτώ ε, μήπως θα πρέπει να έχουμε το θέμα της ρήτρα της ε, δημόσιας τάξης ή ε, κάτι για την δικαιοδοσία όπως ισχύει στις Βρυξέλλες 2. Εκεί υπάρχει ρήτρα ε, και με βάση και τον κανονισμό ε, Ρώμη 3. Η η υιοθέτηση της ρήτρας δημόσιας τάξης θα επέτρεπε στο κράτος μέλος καταρχήν να διαφυλάξει την παράδοση του, την νομική παράδοση, την παραδοσιακή προσέγγιση σε θέματα οικογενειακού δικαίου που όπως ξέρουμε διαφέρει αυτή η νομική παράδοση από χώρα σε χώρα και επίσης θα επέτρεπε στο κράτος μέλος να επισημάνει την ουσία της ε, λειτουργίας της αρχής της επικορικότητας. Αυτή λοιπόν είναι η πρότασή μου ω προ τη συμπερίληψη τη δημόσια τάξη. Τώρα, το δεύτερο τμήμα τη έκθεσή μου έχει μη νομοθετικό χαρακτήρα και ασχολείται με άλλε πτυχές των προβλημάτων των διεθνών υιοθεσιών. Σε αυτό το μη νομοθετικό τμήμα θα έχω διάφορες ε, υποκατηγορίες. Οι βασικές αρχές, η ε, βασική προσέγγιση που ανέφερα προηγουμένως είναι ανδιαφυσβήτητη. Δηλαδή, το θεμελιώδες στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε δράση και την νομοθετική και θα πρέπει να μας ε, καθοδηγεί σε θέματα των παιδιών είναι το συμφέρον του παιδιού, το καλό του παιδιού. Αυτό είναι ο μύθος Αριάδνης και νομίζω ότι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ζητούμενο είναι το συμφέρον του παιδιού, το καλό του παιδιού. Και ο θεσμός της υιοθεσία ακριβώς γι' αυτό θεσπίστηκε προκειμένου να εξασφαλίσει κατάλληλου όρους για τη ζωή και την ευημερία του παιδιού. Και αυτό φυσικά θα πρέπει να μας καθοδηγήσουν, γιατί πρόκειται για παιδιά που δεν μπορούν να ζήσουν ή να αναπτυχθούν σωστά στην βιολογική τους οικογένεια. Αυτό βέβαια είναι δύσκολο κανείς να το αποδεχθεί και μερικές φορές είναι σημαντικό εμπόδιο στο δρόμο της σωστής ανάπτυξης των παιδιών. Αυτή η αδυναμία έβρεση κατάλληλων όρων στη βιολογική οικογένεια και γι' αυτό ανακύπτει η ανάγκη της, νομοθεσ... Θα πρέπει φυσικά κάθε εξέταση να γίνεται περιπτωσιολογικά, εξατομικευμένα. Γιατί το παιδί δεν είναι κτήμα κανενός, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Το παιδί είναι πρόσωπο, είναι άνθρωπος και ως τέτοιο πρόσωπο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Είναι αδύνατο να ε, ε, διανοηθούμε ότι ένα παιδί θα στερήσει τη δυνατότητα ε, να πει τη γνώμη του, να γίνει ακρόαση μαζί του για να ληφθεί υπόψη το συμφέρον του. Και ένα παιδί που μπορεί να είναι μικρό ή να μην αντιλαμβάνεται πολλά θέματα και να μπορεί να εκφραστεί με λόγια, μπορεί να εκφράσει τις ανάγκες του με τη συμπεριφορά του και αυτή τη συμπεριφορά μπορούμε να την παρατηρήσουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην διαδικασία της υιοθεσία. Πιστεύω επίσης ότι σημαντικό είναι το θέμα ε, ο, ο τόπος της ε, ε, διαμονής να μην ε, θεωρηθεί ως ανώτερο αγαθό από τους δεσμούς του αίματος. Γιατί ένα παιδί που χάνει τους γονείς του για τον αλφαβητό λόγο, είτε έχασαν τη ζωή τους, είτε βρίσκονται στη φυλακή και βρίσκονται σε και βρέθηκε σε άλλη χώρα, αλλά στην πατρίδα του βρίσκονται οι παππούδες του για παράδειγμα ή άλλοι συγγενείς του, άνθρωποι που είναι σε θέση να υιοθετήσουν το παιδί και αυτό το θέμα των θεσμών, των δεσμών συγγνώμη, του αίματος θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι ανώτεροι η δεσμοί του αίματος από τον τόπο διαμονής. Και φυσικά, αν μπορούμε να κρατήσουμε τα παιδιά στην πατρίδα μα, είναι σημαντικό για να μην χάνουμε τα νέα ταλέντα. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, το υπέρτατο αγαθό και το ζητούμενο είναι το καλό του παιδιού, το συμφέρον του παιδιού. Και αυτό θα πρέπει να είναι ο βασικό λόγο με βάση τον οποίο θα κρίνουμε οτιδήποτε σε σχέση με την υιοθεσία. Επίση, δεν μπορούμε να δίνουμε ένα παιδί σε υιοθεσία αν δεν κρίνουμε ότι ε, οι βιολογικοί γονείς έχουν χάσει αμετάκλητα το δικαίωμα σε, στην κυδαιμονία του παιδιού. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις μερικές φορές. Άλλα θέματα αφορούν ε, τη λειτουργία του συστήματος ε, που θεσπίζει η Σύμβαση της Χάγης του 1993 σε σχέση με τα δικαιώματα των παιδιών σε περίπτωση διεθνούς νομοθεσίας, ε, υιοθεσίας, συγγνώμη. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η Σύμβαση της Χάγης που σήμερα ισχύει στις περισσότερες χώρες του κόσμου και είναι ενδιαφέρον να μάθουμε και τις εμπειρίες ε, και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης. Και όλες αυτές τις εμπειρίες ε, να τις ε, αξιοποιήσουμε και στις δικές μας ε, νομοθετικές δραστηριότητες. Επίσης να αξιοποιήσουμε και τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Γιατί μερικές φορές το αμελούμε και αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε πώς συνεργάζονται και να συνεργάζονται ε, τα διάφορα θεσμικά όργανα που ασχολούνται με τα δικαιώματα των παιδιών, ή ε, επόπτες, ή ε, συνήγοροι των δικαιωμάτων του παιδιού ή οποιασδήποτε αρμόδιες αρχές ή φορείς αρμόδιοι για τα θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού. Ή επίσης και το θέμα της κατάρτισης των δικαστών που, ή των δικαστικών που εξετάσαμε σήμερα. Είναι σημαντικό οι επαγγελματίες στα θέματα της δικαιοσύνης να είναι καλά καταρτισμένοι και να γνωρίζουν τους ε, κανόνες που ισχύουν για την υιοθεσία στα κράτη-μέλη. Από όλα αυτά που σας είπα, θα σεβεράνατε ότι ο τίτλος της έκθεσης δεν αντανακλά πλήρως το περιεχόμενό της, γιατί αναφέρει ο τίτλος στην διασυνοριακή αναγνώριση της υιοθεσίας, των υιοθεσιών. Και εγώ σας ε, παρήθμισα μια σειρά νέων στοιχείων. Θα έλεγα λοιπόν να τροποποιήσουμε κάπως το τίτλο και να πούμε διασυνοριακές πτυχές των υιοθεσιών. Αυτό θα το προτείνω και αύριο στη συνεδρίαση των συντονιστών. Να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε τον τίτλο της έκθεσης ώστε να αντανακλά καλύτερα το περιεχόμενό της. Και φυσικά Είμαι συνεργάσιμος, ε, διαλλακτικός και περιμένω τα σχόλια της απόψης και των σχεδόν εισηγητών αλλά και των συναδέρφων που ενδιαφέρονται για το ιδιαίτερος ε, ενδιαφέρον αυτό ζήτημα. Θα ήθελα ε, να ολοκληρώσω το έγγραφο τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, αλλά η επίσημη παρουσίαση θα γίνει μάλλον το Μάιο γιατί δυστυχώς τον Απρίλιο δεν θα είμαι παρόν στις ε, συνεδριάσεις της Επιτροπής εξαιτία ε, αποστολών και αντιπροσωπιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα μεταβούν αλλού. Πάντως θα ήθελα, αν γίνεται, να διεκπαιρεώσουμε το θέμα και να ψηφίσουμε πριν τις θερινές διακοπές. Και αυτό θα κρίνει και το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα να έχουμε σχετικά σύντομη προθεσμία για τις τροπολογίες ε, και για την εξέταση τροπολογιών, ώστε Όσο ε, νωρίτερα μπορώ θα υποβάλω το έγγραφο για να ξεκινήσουμε την διορία για τις να τις εξετάσουμε και ενδεχομένω πριν τι θερινές διακοπέ να διεκπαιρεώσουμε το ζήτημα με την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Buddha. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπούντα. Ο κύριος Μπούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο για την παρουσίασή του δεν τον ζηλεύω για όλη αυτή τη δουλειά. Γιατί είναι πράγματι πολύ περίπλοκο το ζήτημα. Από τη στιγμή που μιλάμε για παιδιά και για υιοθεσίε. Θα πρέπει να προτεύσει το συμφέρον του παιδιού πάντοτε στην περίπτωση της υιοθεσία. Και να καταλάβουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι ε, υπερτερεί το απόλυτο συμφέρον του παιδιού. Τι σημαίνει αυτό, να έχει μια στέχη πάνω από το κεφάλι του, να έχει μέσα για να ζήσει. Μπορεί να σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα και ανησυχώ με την έννοια ε, που θα δώσουμε, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε για παιδιά που υιοθετούνται από οικογένειες που δεν αποτελούνται από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Στην Ρουμανία ο γάμος των ομοφιλοφίλων δεν είναι αναγνωρισμένος. Επομένως, είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορούμε να ε, ε, διαβούμε. Πώς θα καθορίσουμε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Σε ορισμένες χώρες η οικογένεια έχει συγκεκριμένο ορισμό στην ένωμη τάξη της εκάστοτε χώρας και υιοθετείται παιδί αναλόγως. Υπάρχουν χώρες όπου ο γάμος των ομοφυλοφίλων επιτρέπεται και μπορεί λοιπόν ένα ζευγάρι να υιοθετήσει τέτοιο παιδί στο διαζύγιο που θα πάει. Θα ανατεθεί επιμέλεια σε έναν από τους δύο γονείς ή σε άλλο ζευγάρι. Θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αυτή η κατάσταση. Είναι υψηλής προτεραιότητας και να προβλεφθούν μηχανισμοί για να καλυφθούν οι εξελίξεις σε όλες τις χώρες, για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την εξέλιξη του παιδιού ε, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υιοθεσία και πριν την υιοθεσία και στην υιοθεσία αλλά και το τι συμβαίνει μετά την υιοθεσία. Ακριβώς για να πούμε ότι ε, σεβόμαστε το ε, συμφέρον του παιδιού. Ε, θα έχω, έχω πολλά να πω για το θέμα αυτό. Στη Ρουμανία είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται εκτενώς σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ για το κείμενο που παρουσιάσατε. Ο Πρόεδρος. Και εγώ η κυρία Ροζιέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το επενθύμισε και ο εισηγητής, είναι πολύ δύσκολες αυτές οι καταστάσεις, οι οικογενειακές, που είναι διασυνοριακές και τα μέσα ενημέρωση έχουν ασχοληθεί και η Επιτροπή Αναφορών και το εργαστήριο το, που οργανώθηκε πρόσφατα, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν πολλές και διαφορετικές πραγματικότητες με πολλές δυσκολίες. Και στα κράτη-μέλη η κατάσταση είναι εξαιρετικά διαφορετική από τη μία χώρα στην άλλη. Αυτό είναι ο λόγος. Επομένως, έχοντας κάνει αυτή τη διαπίστωση, εκφράζω την επιθυμία διεύρυνσης του πεδίου στο οποίο παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε αυτό και μπορούν έτσι να λυθούν γόρδιοι δεσμοί που είναι εξαιρετικά οδυνηροί, με συνέπειες οδυνηρές καθημερινά στην οικογένεια. Υπ' αυτή την έννοια, νομοθετική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι το ευκταίο, το επιθυμητό, πρώτον για να προστατεύσουμε καλύτερα τα παιδιά, που πρέπει να είναι πρώτο μας μέλημα, να αποφύγουμε ε, διακίνηση και να πάμε σε διεθνείς συμβάσεις μόνο εάν άλλες λύσεις δεν προβλέπεται. Χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή δικαστική και νομική. Εγκρίνουμε τη σύμβαση της Χάγης που ε, αυτό είναι μια διασυνοριακή πράξη όμως μια υιοθεσία δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από την άλλη χώρα, δεν έχουμε ίδια μεταχείριση, δεν επιφυλάσσουμε ίδια μεταχείριση σε αυτό. Είναι κάπως περίεργο το ένα και το άλλο. Θα πρέπει να υπάρχουν εγγυήσεις που υπάρχουν στη Σύμβαση της Χάγης να επιβεβαιώσουμε ότι το απότατο συμφέρον του παιδιού και τα θεμελιώδη δικαιώματα του παιδιού επικρατούν και υπερτερούν έναντι οποιασδήποτε άλλη πρόβλεψης και να έχουμε ελάχιστες προϋποθέσεις για τη συνένεση, για τη συγκατάθεση, για τις ε, ιδιότητες ε, των γονιών που υιοθετούν, για τις συνθήκε με τις οποίες λειτουργούν τα ιδρύματα που διαχειρίζονται την υιοθεσία και για να αποφύγουμε τον ε, ε, κερδοσκοπικό χαρακτήρα βεβαίως και εις πρακτικό που θα πρέπει να είναι πλήρως αποκλεισμένος και να μην υφίσταται. Προφανώς κάθε κράτος μέλος επιθυμεί να διατηρήσει τα δικαιώματά του, δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Δεν θα πρέπει ποτέ να αφισβητήσουμε τη σχέση συγγένειας, ούτως ή άλλως θα μπορούσαμε να πάμε στη συστηματική αναγνώριση και στα ε, υιοθεσιών, αναγνώριση υιοθεσιών και δικαιωμάτων που έχουν χορηγήσει τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό θα βοηθήσει τους συμπολίτε μας οι οποίοι πλήττονται από την αποσία αναγνώρισης, πλήττονται από αυτή τη δυσλειτουργία αναγνώρισης των υιοθεσιών σε άλλες ε, χώρες μέλη. Ενθαρρύνω τον εισηγητή ε, στο έργο αυτό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριο Σεραγεφ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά ε, που έχει κάνει σε αυτό το θέμα το τόσο δύσκολο. Πράγματι πιστεύω ότι θα πετύχουμε σημείο ισορροπίας μεταξύ των νομικών πτυχών και των, του ανθρώπινου στοιχείου. Και πράγματι το καλύτερο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί κανείς να υιοθετήσει παιδιά χωρίς τη συγκατάθεση του βιολογικού γονέα. Και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, καταβάλλεται προσπάθεια να επιταχυνθεί η υιοθετική διαδικασία και να αυξηθεί ο αριθμός των παιδιών που δίδονται προς υιοθεσία χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών γονέων. Το 95% των 5.050 υιοθεσιών πέρσι στο Ηνωμένο Βασίλειο έγιναν χωρίς τη συγκατάθεση των βιολογικών γονέων. Και αυτή είναι μια πρακτική διαστροφική θα έλεγα γιατί προσελκύει επιχειρήσεις κερδοσκοπικές που έχουν συμφέρον το κέρδος και αυτό δεν μπορεί να είναι προς όφελος και προς το συμφέρον των παιδιών. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι εξαιρετικά σημαντικό εν ώψη της επικείμενης πρότασης για την, τροπολογία, ε, για την τροποποίηση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α. Πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα για να βελτιώσουμε τη μοίρα, αν θέλετε, τόσο πολλών παιδιών και οικογενειών τους. Στην αναγνώριση των διασυνοριακών υιοθεσιών, το πρωτεύον θα είναι, το πιο σημαντικό, θα είναι να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ κρατών μελών. Επομένως, θα μοιράζονται πληροφορίες και θα συνεργάζονται οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών βάσει άρθρου 55 και 56 και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση ε, της διασυνοριακής ε, υιοθεσίας. Και στο θέμα της κατοικίας του παιδιού, ε, το άρθρο 15, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όλοι θέλουμε να προφυλάξουμε το συμφέρον του παιδιού και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε προτίμηση στις υιοθεσίες μεταξύ της διευρυμένης οικογένειας, οικογένειας του παιδιού, έστω και αν είναι εκτός τόπου κατοικίας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για τα βρέφη. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελούκα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον ε, κύριο Σβιάσκα για την παρουσίαση αυτής της μελλοντικής έκθεσης και να πω ότι το πρόβλημα έλλειψης αναγνώρισης των διασυνοριακών υιοθεσιών μεταξύ των κρατών μελών είναι όντως ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζει η Κομισιόν. Θα ήθελα να πω ότι ήδη από το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης οργάνωσε μια κοινή διάσκεψη στο Στρασβούργο με τίτλο «Προκλήσεις στις διαδικασίες υιοθεσία στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας την ευημερία του παιδιού». Και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν σε αυτή την διάσκεψη ήταν ακριβώς ε, τα προβλήματα που υπάρχουν για τους Ευρωπαίους πολίτες όταν ε, η, υιοθέτηση που, η υιοθεσία που έκαναν σε ένα κράτος μέλος δεν αναγνωρίζεται σε ένα άλλο. Και βεβαίως αυτό οδηγεί σε προβλήματα σε ό,τι αφορά την ελευθερία διακίνησης των πολιτών και στο δικαίωμα του παιδιού να έχει κάποιο πολιτικό έτσι, καθεστώς. Τότε βεβαίως δεν υπήρχε ε, ομόφωνη άποψη για κάποια νομοθετική πρωτοβουλία που θα σχετίζεται άμεσα με τις ε, υιοθεσίε. Και μετά το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δημοσίευσε την Πράσινη Βίβλο για την ελεύθερη διακίνηση των δημοσίων εγγράφων και την αναγνώριση ε, των μητρών. οικογενειακής κατάστασης. Ε, για να μπορεί λοιπόν να αναγνωρίζεται η απόφαση όταν λαμβάνεται στο ένα κράτος μέλος από τα ε, υπόλοιπα. Επίσης, τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησε μια πρωτοβουλία που σχετιζόταν με την ελεύθερη διακίνηση των δημοσίων εγγράφων. Θα θυμάστε ότι ο τελευταίος ε, κανονισμός δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη μετά από πολύ σκληρές συζητήσεις με τα κράτη-μέλη. Ε, ελπίζουμε ότι θα γίνει και αυτό σύντομα. Η Κομισιόν επίσης θα ξεκινήσει τις εργασίες της σε ό,τι αφορά τα έγγραφα οικογενειακής κατάστασης. Είναι ε, καλό βεβαίω να μιλήσουμε τώρα και για το χρονισμό και για την, ε, το πεδίο εφαρμογή αυτή τη μελλοντική πρόταση, αλλά αυτό που θα έχει ω θέμα είναι η αναγνώριση από ένα κράτο μέλο της, των ε, συνεπειών ε, ενός δημοσίου εγγράφου που έχει δημοσιευθεί, εκδοθεί σε ένα άλλο κρατός μέλος και αφορά στην ε, αστική οικογενειακή κατάσταση και των παιδιών που, είναι, που έχουν τύχη Τώρα, σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί σε κράτη-μέλη, μπορούμε να πούμε ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα σε σχέση με περιπτώσεις έλλειψης αναγνώρισης ε, διασυνοριακής υιοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλλον έχουν έρθει στην ε, προσοχή μας κάποιες τέτοιες υποθέσεις, προφανώς θα υπάρχουν και άλλες, αλλά τα κράτη-μέλη δεν διατηρούν στατιστικά στοιχεία και ε, σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν τα διατηρούν, δεν τα μοιράζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η υιοθεσία μειώνεται στην Ευρώπη. Είναι πολύ μικρά τα νούμερα ε, περιπτώσεων υιοθεσιών μεταξύ κρατών μελών. Οπότε το πρόβλημα που έχουμε αφορά στην έλλειψη αναγνώρισης μιας εθνικής υιοθεσίας σε άλλο κράτος μέλος, γιατί προφανώς δεν υπάρχει εναρμόνιση της νομοθεσίας στον τομέα αυτό. Ε, μετά και το ε, εργαστήριο που ανέφερε και ο κύριος Σβιεύσκα, ο εκπρόσωπος της Σύμβασης της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές μίλησε για μια πιθανή σύμβαση για το θέμα αυτό, αλλά Νομίζω ότι αυτό το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό ακριβώς λόγω και του ιδιαίτερου πλαισίου στο οποίο βρισκόμαστε γιατί εδώ μιλούμε για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλο είναι τώρα να αναγνωρίσουμε μια υιοθεσία που έγινε στην Κίνα για παράδειγμα. Είναι τελείως διαφορετικό. Όλα τα κρατημέλη ωστόσο είναι μέρη της σύμβασης του 1993 για, την, ε, για τις ε, διακριτικές υιοθεσίες και όπως αναφέρθηκε η αναγνώριση μιας υιοθεσία η οποία έχει γίνει στα πλαίσια της σύμβασης αναγνωρίζεται ε, δυνάμει του, της νομοθεσίας. Οπότε ας πούμε ότι είναι αυτόματη η αναγνώριση αυτή. Μετά θα Πρέπει να δούμε αν στη μελλοντική πρόταση που έχει να κάνει με την αστική οικογενειακή κατάσταση και τα σχετικά έγγραφα θα μπορούσε η οθεσία να ε, αποτελέσει αντικείμενο ή αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα σχετικά αυτόματο όπως αυτό που απορρέει από τη Σύμβαση του 93. Και για να κλείσω, να πω ότι στον κανονισμό Βρυξέλλες 2α η υιοθεσία εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Εκπίπτει. Οπότε στην ε, μελλοντική αναδιατύπωση δεν ε, νομίζω ότι το θέμα της ε, υιοθέτηση θα μπει ή θα λυθεί μέσω αυτής. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βιέφκα, με προσθέτει το λόγο. Ευχαριστώ επιγραμματικά. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τις ε, παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας, από τα οποία προκύπτει ε, φανώς ότι το θέμα είναι τόσο σημαντικό που καλό θα ήταν να τραβήξει την προσοχή μας ε, και φάνηκε και η περιπλοκότητα του ζητήματος αυτού. Κάτι που αυξάνει και τις δυσκολίες της κατάρτισης της έκθεσης. Πάντως ευελπιστώ ότι θα φέρουμε σε αίσιο πέρα στη διαδικασία. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για την εκδήλωση του ενδιαφέροντος και για τη συνεργασία τους. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε και το σημείο 7 και περνάμε στο σημείο 8 την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα την εκπροσώπηση των εργαζομένων σε ε, διοικητικά συμβούλια στην Ευρώπη. Ο κύριο Γκάσμπαρα Ενρίκο είναι ο συγκεκριτής μα. ο συντάκτη τη γνωμοδότησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχετε το σχέδιο γνωμοδότησης, ε, το οποίο έχω συντάξει και κάποιο καιρό. αποφασίσαμε να το αναβάλουμε για να περιμένουμε την, ε, το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής Απασχόλησης και ε, μας είπαν ότι θα τη λάβουμε τη σχετική έκθεση σχετικά σύντομα. Όπως ε, έχω ξαναπεί, ευχαρίστως θα ακούσω προτάσεις ή σχόλια. Το σχέδιο έκθεσης, έτσι όπως έχει Προς το παρόν βασίζεται στο άρθρο 153 της Συνθήκης της Λισαβόνας και της απορρέουσες διατάξεις. Προς το παρόν 18 κράτη-μέλη έχουν αναγνωρίσει κάποια μορφή συμμετοχής, διαβούλευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων στην εθνική τους νομοθεσία. νομίζω όμως ότι είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να έχουμε πλήρη εναρμόνιση αυτή της νομοθεσία. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ακριβώς η νομοθεσία των πρώτων μελών είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ διαφορετική και λόγω της αρχής της επικουρικότητας θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Θα μπορούσαμε όμως να εκμεταλλευτούμε το ότι υπάρχει και οικονομική κρίση ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ορίσουμε ίσως κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα μπορούσε κανείς να συμμεριστεί σε όλα τα κράτη-μέλη. Προσπάθησα να επικεντρωθώ σε κάποια σημεία τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριλαμβάνονται στην ε, γνωμοδότησή μας. Καταρχάς το θέμα της συμμετοχής, της διαβούλευσης και της ενημέρωσης είναι σημαντικό. Δεύτερον, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που πρέπει να είναι υποχρεωτικοί, το θέμα του ιδιωτικού τομέα επίσης, κατά πόσο αυτό μπορούμε να το ε, διευρύνουμε και για τις ε, ΔΕΚΟ. Τρίτον, να υπάρχει σωστή εκπροσώπηση σε ό,τι αφορά το φύλλο στα διοικητικά συμβούλια και το πέμπτο σημείο είναι να υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση των εργαζομένων στα διοικητικά συμβούλια και βεβαίως να υπάρχουν σωστές διαδικασίες για να εκλέγονται οι εκπρόσωποι των εργαζομένων. Και για τις πολυεθνικές εταιρείες Ευρω... Βεβαίω ε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, αντίστοιχοι κανόνε, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για εταιρείε που ε, υιοθέτουν συγκεκριμένα μέτρα προ όφελο των εργαζομένων μετά από διαβούλευση μαζί του. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από την δουλειά που έχω κάνει για τούτη την έκθεση. Είχα την ευκαιρία να τη συζητήσω με κάποιου συναδέλφου. Ευχαρίστω να ακούσω τι προτάσει σα εφόσον υπάρχουν δεν ξέρω πότε σκοπεύει ο πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης να υποβάλει τη δική του έκθεση σχετικά. Αλλά νομίζω ότι μόλις γίνει αυτό, αυτή τη στιγμή γίνει αυτό, θα μπορέσουμε και εμείς να υποβάλουμε επιπλέον τροπολογίες. Καλό θα ήταν λοιπόν να συντονίσουμε τις εργασίες μας έτσι ώστε να, είμαστε να είμαστε μέσα στα σωστά χρονικά όρια και η δική μας έκθεση να μπορεί να συνταχθεί με την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούντα θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ θερμά τον συντάκτη της νομοδότησής μας για τη μεγάλη διαλλακτικότητα που επιδεικνύει. διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη, τα 28 κράτη-μέλη δεν έχουν ενιαία προσέγγιση για το θέμα αυτό. 18 μόνο από τα 28 κράτη-μέλη έχουν σχετική νομοθεσία. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη και τις ε, μελέτες που έχει πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο ε, Συνδικάτων και θεωρώ ότι θα πρέπει να θεσπίσουμε κάποιους ελάχιστους κανόνες που να εξασφαλίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων ε, και μισθωτών ε, για διαβούλευση και ενημέρωση. Μάλιστα θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων ε, στις οποίες εργάζονται. Και θα πρέπει επίσης κάθε εργαζόμενος να μπορεί να κάνει την επιλογή του, λαμβάνοντας υπόψη την, ε, το δικαίωμά του να ενημερώνεται για τις εξελίξεις της εταιρείας στην οποία εργάζεται, της επιχείρησης. Δεν βλέπω άλλο κανένα ζητάει το λόγο. Δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να σχολιάσει κάτι. Όχι από ό,τι φαίνεται. Οπότε δεν ξέρω κύριε Γκαζμπάρα, θέλετε να δευτερολογήσετε, να σχολιάσετε μήπω αυτά που είπε ο κύριο Μπούντα. Όχι, οπότε ολοκληρώνουμε και το σημείο 8. Μια στιγμή να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Μπούντα και του λοιπούς συναδέλφου γιατί πιστεύω θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μα και με τι τροπολογίε ε, θα διευκρινίσουμε ακόμη καλύτερα τα επιμέρους ζητήματα. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ερωτών ε, είναι παρόντες οι δόκτωρ ε, Πάπετα και Μπόνα. Πάπετας και Μπόνα. Έχουν έρθει οι δύο καλεσμένοι μας. Δεν έχουν έρθει ακόμη οι εμπειρογνώμονες μας για το σημείο 9, οπότε θα κάνουμε ένα διάλειμμα μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Uh, dear colleagues, I think we can... Συνάδελφοι, μπορούμε να ξαναρχίσουμε. Περνάμε στο σημείο 9 που προβλέπει η παρουσίαση των προκαταρκτικών πορισμάτων της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας και της σχετικής αξιολόγησης για τις προθεσμίες στα τροχαία ατυχήματα. Η συγκεκριτής είναι ο υποφαινόμενος θα ήθελα να σας πω ότι συνεχίζουμε το έργο που ξεκίνησε την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία από την ε, κυρία Νταϊόνα Γουόλη, στην οποία ε, οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Και μάλιστα ε, η σχετική διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μελέτη επιπτώσεων ξεκίνησε μια μελέτη για την ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στα τροχαία ατυχήματα και στα θέματα των προθεσμιών. Η Dr. Τζένι Παπέτας και ο Dr. Μάρκο Μπόνα από τη Σκόλα Φορένσε, έγκυροι εμπειρογνώμονες και οι δύο στα θέματα διεθνών τροχαίων ατυχημάτων και αξιώσεων ε, για σωματικές βλάβες από τέτοια ατυχήματα, είναι επικεφαλής ε, της μελέτης ε, ε, για την ανέβριση της προστιθέμενης αξίας ε, της εναρμόνισης των προθεσμιών ε, για τις αξιώσεις που γίνονται από θύματα σε διεθνή τροχιά ατυχήματα. Οι προθεσμίες αυτές διαφέρουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μάλιστα οι διαφορές αυτές οφείλουν, οδηγούν ακόμη και στην απώλεια του δικαιώματος έγερσης αξίωσης ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις διαφορές για τα δικαιώματα των παιδιών, για την έναρξη της προθεσμίας, αναστολή, διακοπή της προθεσμίας ή τα θέματα ανθρώπων με αναπηρίες ε, έχουν τέτοιες διαφορές που διαστρεβλώνουν την άσκηση των ε, δικαιωμάτων. Επίσης, ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο. Συνήθως είναι το δίκαιο του κράτους το οποίο λαμβάνει η χώρα το ατύχημα. Το άρθρο 15 της Σύμβασης Ρωμιδίου προβλέπει κάτι τέτοιο. Επίσης, οι εθνικές διατάξεις για τις προθεσμίες παραγραφής μπορεί να είναι πολύ περίπλοκες και τα θύματα μπορεί να μην είναι εξοικειωμένα με, με τους ε, κανόνες της χώρας στην οποία ταξιδεύουν και στην οποία έτυχε να έχουν το δυστύχημα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν πολύ δυσάρεστε και ανεπιθύμητε συνέπειε για τα θύματα, να δημιουργούν ε, περιτά εμπόδια σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση ε, του δικαιώματο αποζημίωσή του και της έγκαιρης τη της απέτησης τους ε, με ένα σχετικά λογικό κόστος δικαστικό. Για να εξετάσουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα, θα δώσω πρώτα το λόγο στον δόκτωρα Κρίστιαν Σάλμ από την Υπηρεσία Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εφόσον είναι παρόν, είναι και κατόπιν στους δύο εμπειρογνώμονές μας. Θα ήθελα να σας θερμοπαρακαλέσω να μην υπερβείτε το δεκάλεπτο έκαστος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μονάδα προστιθέμενης ευρωπαϊκής αξίας ε, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ασχολήθηκε με το θέμα αυτό των βασικών προθεσμιών για τα διεθνή τροφέα, ε, τροχαία ατυχήματα. Προσπαθήσαμε να εξετάσουμε κατά πόσο η εναρμόνιση τέτοιων προθεσμιών στα κράτη-μέλη θα δημιουργήσει προστιθέμενη αξία. Και για να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό, ε, διαιρέσαμε την μελέτη μας σε τρία τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εξετάζουμε την ανάγκη της εναρμόνισης και της ανάληψης νομοθετικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δεύτερο τμήμα ε, εξετάζουμε τι είδου ε, νομοθετική δράση απαιτείται και στο τρίτο τμήμα ποια θα ήταν η προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας νομοθετική δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης, ε, βρήκαμε δύο κορυφαίους εμπειρογνώμονες, ε, τη δόκτωρα Τζένι Παπέτας και τον δόκτωρο Μάρκο Μπόνα. Η κυρία Παπέτας ε, είναι πανεπιστημιακός του Πανεπιστήμιου του Μπέρμιχαμ και ο κύριος Μάρκο Μπόνα είναι δικηγόρος και διδάσκει στη νομική σχολή του Τουρίνου. Είναι και οι δύο έγκυροι εμπειρογνώμονες. Έχουν δημοσιεύσει πολλά άρθρα για τροχαία ατυχήματα με διασυνοριακό χαρακτήρα και θέματα ασφάλισης οχημάτων. Η Τζένι Παπέτας θα μας παρουσιάσει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, τα προκαταρκτικά πορίσματα της μελέτης που έχω συντάξει. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τα προκαταρκτικά μας πορίσματα. Το θέμα των προθεσμιών έχει θεμελιώδη σημασία για την εξασφάλιση τη αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέματα που αφορούν τι προθεσμίε αφορούν την έγερση τη αξίωση και σε μερικά κράτη, αν δεν γίνουν σεβαστέ αυτέ οι προθεσμίε, τότε χάνεται η ικανότητα τη έγερση τη αξίωση. Αυτέ είναι οι κανόνε περί προθεσμιών. Σε άλλα κράτη-μέλη αν δεν τηρείται η προθεσμία, χάνεται και το ίδιο το δικαίωμα της εξέγερσης, επίσης υπάρχουν, της έγερσης της αξίωσης. Επίσης υπάρχουν και κανόνες περί παραγραφής. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, δηλαδή χάνεται το δικαίωμα της έγερσης της αξίωσης. Η μελέτη που ε, διεξεγάγαμε μαζί με τον Δ. Μπόνα αφορά τους κανόνες ε, προθεσμιών και την ανάγκη εναρμόνιση του Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια κατάσταση ιδιαίτερη σημασίας εξαιτία ε, και, ε, και του νομικού και του κοινωνικού της αντικτύπου. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν χώρα σε κράτος μέλο διαφορετικό από το κράτο διαμονή, ισχύουν εδώ και μία δεκαετία. Η οδηγία για την ασφάλεια των ΙΟΤΑΧΗ ε, προβλέπει ότι τα θύματα που επισκέπτονται μια χώρα μπορούν να, ασκήσουν ε, την ε, αγωγή τους ε, κατά το ασφαλιστή του φορέα αποζημίωσης στο δικαστήριο της χώρας διαμονής τους, κατοικίας τους. Έτσι τα θύματα βρίσκονται σε ένα οικείο νομικό περιβάλλον, μπορούν να ασκήσουν την αγωγή στην μητρική τους γλώσσα και υπόκειται σε νομικές διαδικασίες που μπορεί να μην είναι απόλυτα εκεί τους ίδιους, αλλά σίγουρα είναι γνωστές στους νομικούς συμβούλους τους. Ε, το αποτέλεσμα του εφαρμοστέου δικαίου πολύ συχνά ε, προσδιορίζουν ως εφαρμοστέο δίκαιο το δίκαιο της χώρας ε, που έγινε το ατύχημα. Έτσι, τα θύματα αξιοποιούν τη δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή στην πατρίδα τους. Αυτό όμως σημαίνει ότι το δικαστήριο που θα εκδικάσει την απόφαση θα εφαρμόσει αλλοδαπό δίκαιο, με το οποίο δεν είναι εξοικειωμένο. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει και τους άγνωστους για το δικαστήριο κανόνες των προθεσμιών. Αυτό δημιουργεί πολλές δυσκολίες για τους ενάγοντες. Πρώτα απ' όλα και κυρίως αν οι κανόνε των προθεσμιών δεν είναι κατανοητοί, τότε χάνεται τελείως το δικαίωμα έγκριση αξίωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οι κανόνες περί προθεσμιών είναι περίπλοκοι. Αφορούν τη συνολική προθεσμία, το, την έναρξη τη προθεσμία, το πώς και με ποιο τρόπο μπορούν να διακοπεί να ανασταλεί η προθεσμία. Υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τα παιδιά, για τους ανηλίκους, για τις ανάπηρους, για το κατά πόσο υπάρχει διακριτική ευχέρεια του δικαστήριου σε ό,τι αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων και κάθε κράτο μέλο έχει διαφορετικά συστήματα κανόνων για τις προθεσμίες και για τις επιμέρους πτυχές. Κάτι που δημιουργεί ένα μοναδικό ε, νομικό τοπίο που χρήζει ιδιαίτερο γνώσεων. Επίσης είναι πολύ πιο δύσκολο να οργανωθεί μια ε, αγωγή από την αλλοδαπή. Θα πρέπει ε, να βρεθεί κατάλληλος νομικός εκπρόσωπος, ε, να βρεθεί ο ασφαλιστής, να συγκεντρωθούν ε, αποδεικτικά στοιχεία για το αντίχημα, να γίνουν μεταφράσεις των δικογράφων και επίσης δεν υπάρχει εξοικείωση με το νομικό σύστημα και άρα και με τις προθεσίες. Πολλές φορές έτσι ενάγοντες χάνουν τελείως το δικαίωμα να εγείρουν την απέτησή τους και το, μερικές φορές οι συνολικές προθεσμίες είναι πολύ βραχίες ή υπάρχουν αμφιβολίες ή αφησιμίες για το πότε αναστέλλεται ή διακόπτεται μία προθεσμία. Πολύ συχνά ε, δεν απολυεται τελείως το δικαίωμα της αξίωσης, ε, αλλά δημιουργούνται προσκόμματα στην πρόσβαση της δικαιοσύνης εξαιτίας αυτών των διαφορών στις προθεσμίες. Και μάλιστα όταν ισχύει μια προθεσμία λοδαπού δικαίου, Σίγουρα οι νομικοί σύμβουλοι, οι δικηγόροι χρειάζεται να δαπανίσουν πολύ περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν με το δαπό δίκαιο. Κάτι τέτοιο δεν θα χρειαζόταν ήταν το, το δίκαιο του εθνικό του δίκαιο. Κάτι τέτοιο αυξάνει τα δικαστικά έξοδα. Μερικές φορές μπορεί να χρειάζεται και ε, γνωμοδότηση εμπειρογνώμονα ε, από τον τόπο ατυχήματο για να ε, γίνει αντιληπτό πώς λειτουργούν οι προθεσμίες. Όλα αυτά δημιουργούν προσκόμματα, ειδικά θα χρειαστεί συγκέντρωση αποδείξεων από αλλοδαπό εμπειρογνώμονα. Η διαδικασία γίνεται και πιο χρονοβόρα και πιο δαπανηρή. Και επίσης είναι ε, και ψυχολογική η βλάβη για το θύμα που μπορεί να έχει άγχος και αβεβαιότητα για την έκβαση της αξίωσης του. Είναι πολύ περιπλοκή η κατάσταση αυτή και η οδηγία για την ασφάλεια των ΙΟΔΕΧΗ κανονικά έπρεπε να, ε, και στόχο είχε να διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων. Η περιπλοκότητα της κατάστασης και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ανάγοντες ε, δίνει εύλογους λόγους για την ανάγκη εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τις προθεσμίες, τους χρονικούς περιορισμούς. Κάτι τέτοιο δεν είναι καινούριο. Η πιθανότητα εναρμόνιση αυτών των μέτρων ε, ανεφάνει ε, πριν από 15 χρόνια και πρόσφατα είχαμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2009 και δύο δημόσιες διαβουλεύσεις ε, που ακολούθησαν και που έδωσαν δηλαδή για συζήτηση βασικών ε, σενάριων. Τρία από αυτά τα σενάρια λήφθησαν ιδιαίτερη υπόψη, όπως η ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των θυμάτων. Ε, θεωρούμε ότι οι κανόνες περί προθεσμιών ε, χρήζουν ιδιαίτερη ερμηνεία σε κάθε περίπτωση εξαιτία του περίπλοκου χαρακτήρα τους και δεν αρκούν ε, γενικές δηλώσεις για τις πιθανές συνέπειες των προθεσμιών αλλοδαπού δικαίου γενικά και όριστα. Χρειάζεται εξατομικευμένη ανάλυση. Τα απορίσματα μας προβλέπουν ότι η θέσπιση εναρμονισμένης νομοθεσίας θα ήταν ο καλύτερος δρόμος για να λυθούν τα προβλήματα. Επίσης θα πρέπει να καλυφθούν βασικές ε, πτυχές των ε, προθεσμιών όπως έναρξη, ε, διακοπή και αναστολή, ειδικά δικαιώματα των παιδιών ή των ατόμων με αναπηρίες. Επίσης θέμα φορέων αποζημίωσης ή ασφαλιστών και η διασύνδεση με την οδηγία για τις ασφάλειες αυτοκινήτων. Εναρμοσμένοι όρδε κανόνες θα πρέπει να αφορούν μόνο διασυνοριακές καταστάσεις. Τώρα, και στο συμπέρασμα αυτό και στην υποβολή των προτάσεών μας για την εναρμόνιση της νομοθεσίας λάβαμε υπόψη ένα ευρύ φάσμα παραγόντων. Καταρχήν το, την ικανότητα των διαφόρων θεσμικών οργάνων να δούμε βάσει τη συνθήκη, ιδιαίτερα αν είναι κατά πόσο, είναι σωστή και επαρκή μια τέτοια δράση και αν πληρούν διαρχέ επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Όλα αυτά τα θέματα θα αναλυθούν διεξοδικά στην έκθεση που θα ακολουθήσει. Το συμπέρασμα πάντω είναι ότι εφόσον υιοθετείται σωστή προσέγγιση στην εναρμόνιση, θα υπάρξει σωστή νομική βάση με βάση το άρθρο 81 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τι αρχέ ε, τη ε, επικουρικότητα και τη αναλογικότητα που θα τηρούνται. Σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο των εναρμονισμένων κανόνων. Οι υπάρχοντες εναρμονισμένοι κανόνες που που αφορούν τα δικαιώματα των επιβατών, για παράδειγμα, υπάρχουν ήδη. Και πολλά νομοθετικά μέτρα δείχνουν ότι τα δικαιώματα επιβατών για όλα τα μέσα μεταφορά ε, τυχάνουν προστασία ε, και ελάχιστων εγγυήσεων σε ό,τι αφορά του κανόνε για τι προθεσμίε. Κάτι που ε, βελτιώνει την κατάσταση ε, στα μέσα μεταφορά, αλλά και τα διασυνοριακά ατυχήματα δεν υπάρχουν τέτοιε ελάχιστε εγγύησεις. Ούτε υπάρχει ενιαίο μοντέλο που μπορεί να ακολουθηθεί σε περίπτωση εναρμόνιση των ε, κανόνων για τι προθεσμίε. Σε ό,τι αφορά την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά του χρονικού περιορισμού. Η νομολογία δείχνει ότι χρειάζεται ένα ελάχιστο επίπεδο προστασία του δικαιώματο ε, αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και αυτό μπορεί να καταστραγηθεί σε περίπτωση προθεσμίες που καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στο δικαστήριο, είτε γιατί δεν είχε την ευκαιρία ο ενάγων να αξιολογήσει πλήρως τη ζημία ή να βρει τον αυτούργο ε, ή τον ε, υπόλογο ε, της αποζημίωσης και ούτω καθεξής. Οι προτάσεις για, για την εναρμόνιση των προθεσμιών προτείνουν πολλές και διάφορες ε, προτάσεις. Για παράδειγμα, διεξοδικές, ε, ε, διεξοδικές διατάξεις ή πολύ γενικές διατάξεις. Τα προκαταρκτικά προορίσματα δείχνουν ότι γενικές διατάξεις ελάχιστων θεμάτων θα αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα των εναγόντων και κυρίως το δικαίωμα να σταθεί κατά το ασφαλιστή και τηρούν τέτοιε γενικές ε, αρχές περισσότερο τι τις αρχές και αναλογικότητας. Επίσης, ε, διασκεδάζονται οι αμφιβολίες που έχουν ε, αρμόδιο του ασφαλιστικού κλάδου σε ό,τι αφορά την ιδέα της εναρμόνισης. Βέβαια όλα αυτά θα αναφερθούμε λεπτομέρειες στην έκθεση, καθώς και την πιθανή αξία που θα έχει η εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα είναι πολύ σημαντική. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προστιθέμενη αξία, σαφώς υπάρχει προστιθέμενη αξία στη μείωση του χρονικού κόστους αλλά και του ψυχολογικού κόστους σε ό,τι αφορά τη διαφορά των προθεσμιών και την περιπλοκότητα και την αβεβαιότητα που δημιουργούν οι διαφορετικές τις προθεσμίες. Αλλά και σημαντικές οικονομίες χρηματικές θα γίνουν με μια τέτοια εναρμόνιση. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχουμε στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που λαμβάνουν κάθε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για τον αριθμό των αξιώσεων και των αγών που εγείρονται και που δημιουργούν προβλήματα στις προθεσμίες. Πάντως υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για προστιθέμενη αξία της εναρμόνισης. Ε, μάλιστα φαίνεται από στοιχεία ότι 16.000 ευρώ αναξίωση ε, χάνονται κατά μέσο όρο όταν αφορούν προσωπικές, ε, ζημίες, προσωπικές βλάβες και 2.000 ε, για περιουσιακές βλάβες εξαιτία των προθεσμιών. Και βέβαια δεν καλύπτουμε εδώ την περίπτωση τροχαίου, ολέθρη τροχαίου που θα έχει καταστροφικές βλάβες ή ζημίες ε, στα δικαιώματα του ενάγοντος. Επίσης η ανάλυση μας δείχνει ότι περίπου 250.000 ε, άνθρωποι κάθε χρόνο ε, επηρεάζονται από περιτά προσκόμματα σε ό,τι αφορά την έγερση της αγωγής τους. Άνθρωποι δηλαδή που όχι χάνουν μόνο το δικαίωμα άσκησης της ε, απέτησης, αλλά που ε, αντιμετωπίζουν προβλήματα εξαιτία τη εφαρμογή διαφορετικών προθεσμιών. Θεωρούμε ότι το επιπλέον δικαστικό κόστο που σχετίζεται με τι προθεσμίε είναι κατά πάσα πιθανότητα γύρω στα 600 ευρώ ε, ανά αγωγή, ανά απέτηση. Και μάλιστα χρειάζεται και η γνωμοδότηση αλλοδαπού εμπειρογνώμονα για την εφαρμογή των, των προθεσμιών αλλοδαπού δικαίου θα είχαμε επιπλέον ένα 300 ευρώ ανά αγωγή. Και το ε, αναγάγουμε αυτό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σύνολο, βλέπουμε ότι οι δράσεις εναρμόνισης τέτοιων προθεσμιών θα μπορούσαν να μας εξοικονομήσουν κάθε χρόνο μέχρι και 300 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα το ποσό αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το σε συναφές ε, ε, δικαστικό κόστος, τα, τα τέλη εμ, για συμπληρωματική μετάφραση, γιατί δεν υπάρχουν λεπτομεριακά στοιχεία και έτσι αυτά τα έξοδα δεν τα λάβαμε καν υπόψη. Εν κατακλείδη, η απόφαση εναρμόνισης των κανόνων χρονικού περιορισμού ή προθεσμιών για άλλες αξιώσεις που ε, προκύπτουν από μέσα μεταφοράς ε, δεν εξαρτάται από την ανάγκη του να δείξουμε αν κάποιο ε, επωφελείται από μια τέτοια δράση ή αν έχουν γίνει αρκετέ οικονομίε. Αλλά με την πρόθεση τη ελεύθερη διακίνηση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε αρκετού λόγου για να ταχθούν υπέρ τη εναρμόνιση των χρονικών περιορισμών για διασυνοριακά τροχαία ατυχήματα. Βέβαια η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη ε, και σίγουρα με την εναρμόνιση θα γίνουν πολλές ε, οικονομίες. Σας ευχαριστώ. Ε, thank you very much, Dr. Pepitas. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ο Δόκτωρ Μπόνα δεν είναι εδώ. Σωστά. Κατάλαβα. Ναι δυστυχώς είναι άρρωστος, δεν μπορούσε να παρευρίσκεται σήμερα. Εντάξει, δεν έχω κάποιον το λόγο. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε στην ε, πλήρη σας έκθεση μια απάντηση στο εξής ερώτημα. Σε κάποια κράτη-μέλη το θέμα της ε, περίοδου παραγραφής, της προθεσμίας παραγραφής, ανήκει στο ουσιαστικό δίκαιο. Σε άλλες χώρες στο διαδικαστικό. Αυτό ίσως επηρεάσει την νομική βάση για μελλοντική εναρμόνιση. Μπορεί να περιπλέξει με κάποιο τρόπο τον στόχο αυτό που έχουμε τις εναρμόνισης. Ευχαρίστως να το συμπεριλάβουμε το θέμα αυτό στην έκθεση, αλλά έτσι προκαταστικά να πω ότι δεν νομίζω ότι η νομική βάση θα επηρεαστεί από την επιλογή του δικαίου. Όντως σε κάποια κράτη-μέλη είναι θέμα εισαστικού δικαίου και σε κάποια άλλα όχι. Αλλά αν πάρουμε μια προσέγγιση όπου υπάρχει ένα ελάχιστο πρότυπο εναρμόνισης και μετά επαφείται στο κράτος μέλος ο τρόπος και η μορφή με την οποία θα εφαρμοστεί αυτή η εναρμόνιση, τότε δεν νομίζω ότι, δεν περιμένω δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια επιπλοκή. Θα μπορούσαμε βεβαίω να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο και να συμπεριλάβουμε συγκεκριμένα σχόλια και απαντήσεις στην έκθεση σχετικά. Ευχαριστώ γιατί όντως για χώρες όπως οι δικέ μου θα έπρεπε να υπάρξει αλλαγή στον αστικό μας κώδικα για να μπορέσει να γίνει αυτή η εναρμόνιση. Οπότε καλό θα ήταν να έχουμε μια απάντηση από εσά. Ο κύριο Ράντεφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για την αρχική τους αξιολόγηση μιας ε, πιθανής προσθέμενης αξίας ε, της, ε, όλου αυτού του εγχειρήματος εναρμόνισης της παραγραφής για τα τροχαία ατυχήματα. Αυτό είναι σημαντικό για τους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι καθημερινά έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορες δυσκολίες που προκύπτουν από αυτές ακριβώς τις διαφορετικές προθεσμίες που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Διαφορές που θα μπορούσαν να, να οδηγήσουν σε πολύ άσχημες συνέπειες για τα θύματα των τροχιών ατυχημάτων και να τους δημιουργήσουν επιπλέον εμπόδια όταν προσπαθούν να γύρουν την αξίωσή τους σε κάποιο άλλο κράτος μέλος σε σχέση με αυτό στο οποίο κατοικούν. Και μπορεί να χάσουν ακόμη και το δικαίωμα έγερσης τη αξίωσή του. Η ε, μικρότερη βεβαίω προθεσμία ενό κρατου μέλου, αν ένα κράτο μέλο υποβάλλει δηλαδή μικρότερη ε, προθεσμία, θα μπορούσε ίσω να ε, αποζημιωθεί μέσω μια πιο γρήγορη ταχεία διαδικασία εφαρμογής των κανόνων. Είναι δύσκολο βεβαίω ποιο να, καταλάβει κανεί ποιο θα πρέπει να είναι το συνολικό πλαίσιο, αλλά παρόλα αυτά η καθοδήγηση που δίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση του 2007 θα μπορούσε ίσως να φανεί χρήσιμη. Υπάρχει ανάγκη να υπάρξει ευαισθητοποίηση, αύξηση της ευαισθητοποίησης, όχι μόνο όσων, όσον, τους, αφορά, αλλά και όλων των πολιτών για τα θέματα αυτά, γιατί ε, τροχιά ατυχήματα γίνονται παντού. Ε, θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε σε μια λύση η οποία θα βασίζεται στη σύμβαση της ε, Χάγης και στην Ρώμη 2 για το Εφαρμοστείο δίκαιο. Ευχαριστώ. Ε, Delvaux. Η κυρία Ντελβό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση ήθελα να υποβάλω. Έχω δίκιο όταν καταλαβαίνω ότι στα ελάχιστα πρότυπα το πιο σημαντικό είναι η εναρμόνιση της περίοδου κατά τη διάρκεια της οποίας μπορεί κανείς να ασκήσει αγωγή. Βλέπω αυτή την απαρίθμηση. Ποιο είναι το πιο επίγον, ποιο πρέπει να ρυθμίσουμε πρώτα. για να διευκολύνουμε τη ζωή όσων έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Ο κύριος Λεμπρέτον. Και εγώ έχω ένα ερώτημα να απευθύνω. Καταρχάς σας ευχαριστώ που ήρθατε. Πράγματι το ζήτημα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και κάνατε σωστή ανακεφαλαίωση των προβλημάτων. Πράγματι τα τροχιά ατυχήματα είναι δύσκολο να ε, ρυθμιστούν νομικά γιατί υπάρχουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής, διαφορετικές ένομες τάξεις, 250.000 άνθρωποι πλήττονται ετησίως και δυσκολεύονται να αποζημιωθούν. Όλες αυτές οι περιγραφές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, ωστόσο δεν με καλύψατε ως προς τις προτάσεις, παρόλο που είμαστε σε φάση προβληματισμού ακόμα, εσείς υιοθετείτε συγκεκριμένη θέση και είστε υπέρ της εναρμόνισης ε, του χρόνου ε, παραγραφής, της διάρκειας παραγραφής. Για, ποιο, για ποια διάρκεια μιλάμε όμως. Μπορείτε να μας κάνετε μια παρουσίαση πώς έχει η προθεσμία παραγραφή σε κάθε χώρα, σε ορισμένες χώρες τουλάχιστον, για να ξέρουμε προς ε, τα που πηγαίνουμε, να είναι προθεσμία δύο μηνών, τριών μηνών, ε, ποια χώρα την προθεσμία θα ακολουθήσουμε. Προς το παρόν επικρατεί σύγχυση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Παπέτας να απαντήσει. Και εγώ σας ευχαριστώ όντως ε, είναι, ποιες είναι οι πιο σημαντικές ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουμε. Ε, εσείς ρωτάτε ποιο είναι το πιο σημαντικό στην πρώτη σας ερώτηση. Δεν είναι τόσο σαφές. Ίσως δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει να τρέχει αυτή η προθεσμία μπορεί κανεί να την έχει αναστείλει ενώ τελικά δεν, το έχει καταφέρει γιατί ο τρόπο με τον οποίο αναστέλλεται μια προθεσμία στο ένα κράτο μέλο είναι διαφορετικό με τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο πράγμα γίνεται σε άλλο κράτο μέλο. Έχουμε παραδείγματα περιπτώσεων όπου τα άτομα θεώρησαν ότι είναι μέσα στην προθεσμία ενώ τελικά κατάλαβαν ότι δεν είχαν τηρήσει την προθεσμία σύμφωνα με τους ε, εφαρμοστέους κανόνες και υπήρξαν δυσκολίες. Ενδεχομένως να μην έχουν χάσει το δικαίωμα άσκησης αγωγής, αλλά ε, ο, η ασφαλιστική εταιρεία του ε, διάδικου μέρους μπορεί να ε, δώσει λαβή για επιπρόσθετες δικαστικές διαδικασίες, επιπρόσθετες ακροάσεις και το καθεξής. Επομένως, σε χώρες όπου η προθεσμία είναι σύντομη, το ζήτημα αυτό είναι πολύ ακαθόδες, γιατί χρειάζεται χρόνος να οργανώσει κανείς ε, την άσκηση των ενδίκων μέσων από το εξωτερικό. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πότε και πώς θα αναστέλλεται αυτή η προθεσμία και ε, με ποιους τρόπους θα διακόπτεται δηλαδή και πώς θα μετά θα ξαναξεκινά να συνεχίσει να τρέχει. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Λεμπρετό, πράγματι είναι πολύ διαφορετικές οι χρονικές περίοδοι. Από ένα χρόνο είναι η πιο σύντομη περίοδος, μέχρι και 30 χρόνια η πιο μακρά χρονική περίοδος και όλα τα ενδιάμεσα, όλες οι ενδιάμεσες αποχρώσεις έννοιες υπάρχουν. Και μάλιστα σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν και διαφορετικές προθεσμίες κατά που εξαρτώνται από το κατά πόσο η διεκδίκηση είναι μόνο στο αστικό ή και στο ποινικό σκέλος. Όλα αυτά δεν ε, βοηθούν τον ενάγοντα γιατί χρειάζεται και νομική αξιολόγηση της ε, αγωγής, της διεκδίκησης. Εμείς εξετάσαμε τους εφιστάμενους κανόνες Κάναμε συγκριτική ανάλυση των διαφορετικών ε, περιορισμών στην χρονική ισχύ που ισχύουν στα κράτη-μέλη και εξετάσαμε και τις υφιστάμενες προτάσεις ε, εναρμόνισης. Και το πώς αυτά ισχύουν σε άλλους τρόπους μεταφοράς. Και ως προκαταρκτικό συμπέρασμα έχουμε καταλήξει στο ότι ίσως μια περίοδος τεσσάρων ετών να ήταν κατάλληλη. Προκαταρκτικό βέβαια αυτό το συμπέρασμα και επιδέχεται αλλαγών προφανώς. Δεν ξέρω αν απάντησα το ερώτημά σας κύριε Λεπρετού. Καλώς, ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, αφού δεν θέλει κάποιος άλλο το λόγο, να σας ευχαριστήσω Κύριε Παπέτα για την παρέμβασή σας. Στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλετε το λόγο? Όχι. Βλέπω λοιπόν ότι έχουμε εξαντλήσει την εξέταση της ημερήσιας διάταξης για την πρωινή μας συνεδρίαση. Σας εύχομαι καλή όρεξη. Θα τα πούμε στις 3.